So, liebe αγαπητοί συνάδελφοι στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Είμαστε στο σημείο 15 εσείως και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τον Επίτροπό μας, τον κύριο Τζον Ντάλι, που είναι Επίτροπος για θέματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας τροφίμων. Καλωσορίζω και τη Γενική Διευθύντρια κυρία Τεστόρη και όλο του στο επιτελείο της Γενικής Διεύθυνσης ε, για την οποία στην οποία μάλλον είναι αρμόδιοι για την Επιτροπή μας. Η ασφάλεια τροφίμων, όπως γνωρίζουμε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και λεπτό. Έχουμε περάσει νύχτες ολόκληρες μαζί ε, να συζητούμε και να διαπραγματευόμαστε για το θέμα αυτό. Και πρόσφατα να βάγισε ε, ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα, το novel food, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάνε καλά αλλού τα πράγματα σε άλλα θέματα και άλλους φακέλους που είναι ακόμα στην σε διάταξη επίκυνται. Η δημόσια υγεία είναι μια μεγάλη υπόθεση ε, την οποία παρακολουθούμε πάρα πολύ σοβαρά παρόλο που η Επιτροπή μας είναι ευρύτατη, είναι τόσο μεγάλο το φάσμα των ε, αρμοδιοτήτων και των θεμάτων που μας απασχολούν. Νομίζω γιατί η πολιτική δημόσια υγείας θα έπρεπε να είχαμε περισσότερο χρόνο να αφιερώνουμε. Συναντιόμαστε λοιπόν σήμερα στα πλαίσια του λεγόμενου διαρθρωμένου διαλόγου, γιατί η Συμφωνία Πλαίσιο Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει να ανταλλάσσουμε απόψεις για το σχεδιασμό των διαφόρων τομέων της πολιτικής μας, όπερ και θα γίνει σήμερα και χαίρομαι που ο Επίτροπος μας ενημερώνει συχνά και άτυπα πολλές φορές και θα του δώσω το λόγο για να μας ενημερώσει για τα θέματα που μας απασχολούν και έχουμε μπροστά μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Well, thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ ένα χρόνο περίπου από τότε που ανέλαβα και ένα χρόνο από τότε που πρωτοπευθύνθηκα στην Επιτροπή σας. Με βοήθησαν πάρα πολύ οι συμβουλές και η προσφορά της Επιτροπής Περιβάλλοντος το τελευταίο 12 Προσβλέπω σε μια συνεχιζόμενη επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ μας. Το τελευταίο δωδεκάμινο, κατά την άποψή μου, κατάφερε να ενισχύσει την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Δηλαδή, από κοινού καταφέραμε να ολοκληρώσουμε σημαντικές νομοθετικές διαδικασίες που αφορούν την, την, τη δωρεά οργάνων, την φάρμακο επιφυλακή, τις ε, διαμεθοριακές παθήσεις και άλλα. Βεβαίως θυμόμαστε και την αποτυχία των νέων τροφών, Θυμόμαστε όμως τώρα, ας σκεφτούμε τώρα το πρόγραμμα της Επιτροπής για φέτος και για το 2012 και θα ήθελα να επισημάνω τις γενικές κατευθύνσεις του. Ξεκινώντας από τη μελλοντική πρόταση της Κομισιόν να αναθεωρήσει την οδηγία προϊόντων καπνού που σχεδιάστηκε το 2012. Ο καπνός δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα προϊόντα. Ο καπνός είναι ένα εξαιρετικά εθιστικό και εξαιρετικά τοξικό προϊόν. Κυρίως με απασχολεί το θέμα των νεαρών Ευρωπαίων καπνίζουν εις βάρος της υγεία τους και το μέλλον, του μέλλοντός τους. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που ένας στους τρεις 15χρονους ήδη καπνίζει. Πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή ο καπνός να γίνει λιγότερο ελκυστικός, κυρίως στους νέους και να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος γνωρίζει ακριβώς τι κάνει ο καπνός στην υγεία τους. Τώρα εξετάζω τα νομοθετικά μέσα για να ενισχυθούν οι προειδοποίησεις για την υγεία στα πακέτα και να ε, ρυθμιστούν τα θέματα της, ε, των γεύσεων και των, ε, του καπνού και να μελετήσουμε άλλα προϊόντα όπως τα e-cigarettes. Υπάρχει μέσα σε αυτό το πνεύμα προτίθεμαι να προτείνω μια αναθεώρηση της οδηγίας ε, προϊόντων καπνού στην αρχή του επόμενου έτους και ελπίζω να έχω την υποστήριξη της Επιτροπής σας αλλά και του Κοινοβουλίου συνολικά. Επιπλέον συμμερίζομαι την ανησυχία του Κοινοβουλίου να μάθουμε από την εμπειρία μας την πανδημία του ΙΤΑ 1 και να λάβουμε ανάλογα μέτρα σκοπεύω μέχρι το τέλος του χρόνου να προτείνω ένα πακέτο που θα αφορά τις πανδημίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αναφέρεται στις ε, συνέπειες μιας μεγάλης σειράς απειλών. Έχει ξεκινήσει διαβούλευση μέχρι το τέλος του μήνα επ' αυτού. Όπως θα γνωρίζουν τα μέλη, σκοπεύω να προτείνω αναθεώρηση της οδηγίας κλινικών δοκιμών στο της περίοδου 2010-2012. Η κλινική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται και ο αριθμός αιτήσεων για κλινικές δοκιμές έπεσε κατά 20% από το 2007 έως το 2010 πρέπει να φροντίσουμε η κλινική έρευνα να παραμείνει στην Ευρώπη. Αυτό είναι ζωτική σημασία ε, για τους ε, ασθενείς που πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πιο καινοτόμα θεραπεία κάθε φορά και να υπάρξει υπεροχή στην έρευνα στην Ευρώπη. Η άτυπη διαβούλευση περιλαμβάνει ιδέες για τη βελτίωση των κλινικών ερευνών βελτιωμένη και πιο ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες για τα φάρμακα είναι επίσης σημαντικός στόχος. Κάποιοι ασθενείς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να μάθουν για την πάθησή τους και τις διαθέσιμες εναλλακτικές παθή, ε, για θεραπεία, μεταξύ των οποίων και τα φάρμακα. Πιστεύω ότι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν πληροφορίες αυτές. Επιπλέον, οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αποτελούν φίλτρο ανάμεσα σε αυτούς που κατέχουν την άδεια διακίνησης και εμπορία και στου ασθενεί. Η αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να έχει εγκριθεί μέχρι το Μάιο, θα τροποποιηθεί ανάλογα με ε, την κατεύθυνση αυτή, επί τη βάση αυτής της κατεύθυνσης. Η Ευρώπη έχει καλό θεσμικό πλαίσιο για τις ιατρικές συσκευές, όμως πρέπει να βελτιωθεί για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας των ασθενών και να προωθηθεί καινοτομία. Το 2012 η Κομισιόν θα προτείνει ε, πρόταση αναδιατύπωσης της σχετικής οδηγίας. Τα βασικά στοιχεία συζητήθηκαν τον περασμένο μήνα στην διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την καινοτομία και ε, στην, στον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας, στην οποία συμμετείχε ευγενώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η υγεία των καταναλωτών της Ευρώπης φυσικά εξαρτάται και από τα ασφαλή τρόφιμα. Πράγμα που σημαίνει ότι τα ζώα θα πρέπει να ανατρέφονται και να διατηρούνται με τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Θα πρέπει να ε, ε, θεσπιστεί μια νέα στρατηγική ευζοίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Υπάρχει ένας νέος νόμος της ευζοίας των ζώων Κοινοβούλιο και ε, μελετάμε τις προτάσεις σας. Επιπλέον, η επιπλέον διαδικασία για την περαιτέρω εναρμόνιση έχουν ξεκινήσει. Όπως γνωρίζει η Επιτροπή η Κομισιόν εργάζεται στο θέμα της, ε, του νόμου για την υγεία των ζώων που περιμένουμε μια επίσημη πρόταση του χρόνου. Αυτός θα ψηφιστεί, μάλλον θα στηριχθεί στη βασική αρχή ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Και θα υπογραμμιστεί η, σημασία της υγείας που συνδέει τα ζώα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Φέτος θα ε, ακολουθήσουμε τη συμφωνία του 2010 χάρη στην εμπλοκή της κυρίας Ντεμπρόν με την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα κατοικίδια. Όσον αφορά τα φάρμακα, υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικών κτηνιατρικών φαρμάκων στην Ευρώπη. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει αναθεώρηση σχετικής νομοθεσίας με σκοπό το 2012 να υπάρξει, να εγκριθεί πρόταση που θα προσπαθήσει να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων. Τώρα, όσον αφορά τα τρόφιμα επανεξετάζονται οι επίσημοι έλεγχοι για να απλουστευθεί και να ενοποιηθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση μας. Η αναθεώρηση αυτή θα κοιτάξει το θέμα του ελέγχου, του ελέγχου των κτηνιατρικών φαρμάκων και των εισαγω... ελέγχου του κατά την εισαγωγή. Πρέπει η Κομισιόν, να χρηματοδο... η κοινότητα να χρηματοδοτήσει τις, ε, ε, τις ε, ελεγκτικές αρχές μέσω των τελών που θα εισπράττονται. Και εδώ έχει σχέση και το πακέτο υγιεινής των τροφίμων που δεν σημαίνει αναδιατύπωση όλου του πακέτου, αλλά μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση απλούστευση των διαδικασιών και της αντιμετώπισης των μεταβατικών μέτρων και κυρίως μερικών μέτρων που αφορούν την, τον έλεγχο του κρέατος. Έχει γίνει πρόοδος στον τομέα των εγκεφαλοπαθειών. Βρισκόμαστε σχεδόν στην εξάλληψη της ασθένειας ε, χάρη στην, στα νέα ισχυρά μέτρα. Τώρα, ένα βήμα στον, στον νέο δικό χάρτη των ε, μεταδοτικών εγκεφαλοπαθειών μπορεί να γίνει η Κομισιόν προτείνει να αναθεωρηθεί η μέθοδος ελέγχου των, ε, των βοηδών για μεταδοτικές εγκεφαλοπάθειες και τώρα αυτή η πρόταση έχει γίνει δεκτή υπάρχουν διατάξεις πλήρους απαγόρευσης ε, ζωοτροφών. Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι όλες οι, όλοι οι όροι που στηρίζονται ε, επιστημονικά θα πρέπει να υφίστανται πριν βεβαίως συμφωνήσουμε σε κάποιες τροπολογίες. Προσβλέπω στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτού, ενώ, η οποία υποβλήθηκε από την κυρία Ντάκμα Ροτ Μπέραντ χτες το απόγευμα στην Επιτροπή. Τέλος, το πρόγραμμα εργασίας για το διάστημα 2012 προβλέπει την έγκριση ενός νέου ευρωπαϊκού νόμου για την ε, υγεία των φυτών, για την προστασία της γεωργίας που αφορά και τα ξένα ζυζάνια και τις παθήσεις. Θέλω τώρα να αναφερθώ σε κάποια άλλα θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή. Όσον αφορά την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, έχω ε, παρατηρήσει την έκθεση της κυρία, παρακολουθήσει στενά την έκθεση της κυρίας Λαπάζ και τις προσπάθειες που γίνονται για να ε, μπείτε σε περισσότερες λεπτομέρειες και να δικαιολογήσετε τις παγορεύσεις καλλιέργειας. Οι λόγοι για τους οποίους η Κομισιόν αναφέρθηκε σε αίτια που έχουν σχέση μόνο με την επίπτωση των οργανισμών αυτών στην υγεία και στο περιβάλλον είναι για να μην ε, επέλθει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Πρέπει να προτείνω, να υπογραμμίσω ότι ε, στόχο της Επιτροπής είναι να δω έχουν την δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μην καλλιεργούν. Το θέμα δεν είναι ε, θέμα επιλογής όταν εμπλέκονται κίνδυνοι, είναι θέμα υποχρέωσης και η φυστάμενη νομοθεσία προβλέπει μέτρα περιοριστικά. Το πρωί εγκρίνατε τροπολογία στο σχέδιο έκθεσης και μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να την ευήκονους και να συζητά τις τροπολογίες που, ε, ε, στις απόψεις της Επιτροπής Η Κομισιόν είναι αποφασισμένη να συνεργάζεται στενά με τους συνομοθέτες. Όσον αφορά την πρόταση για τους καταναλωτές και τα τρόφιμα, έκθεση κυρία Σόμερ, φτάνουμε τώρα στην κρίσιμη φάση της νομοθετικής διαδικασίας. Είμαι πεπισμένος ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συμφωνήσουν μεταξύ τους και εγώ είμαι διατεθειμένος να στηρίξω τις προσπάθειες προς μια επιτυχημένη συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Η Κομισιόν στηρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση για την ε, σήμανση στον προστινό μέρος της, συσκευασία για τα πέντε θρεπτικά στοιχεία. Ελπίζω να το επιτύχουμε. Θα υπάρξει με αυτόν τον τρόπο προστασία των καταναλωτών χωρίς να επιβάλλουμε άχρηστα περιτά βάρη στους παρασκευαστές. Θα ήθελα πριν ολοκληρώσω να αναφέρω μια σημαντική πρωτοβουλία που σας ενδιαφέρει ξέρω ιδιαίτερα, ιδίως κάποια από τα μέλη σας. Το ILET είναι η εταιρική σχέση ε, καινοτομίας που είναι η πρώτη τέτοια εταιρική σχέση στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Ε, Στόχος της ε, εταιρικής αυτής σχέσης είναι να αυξηθεί κατά δύο χρόνια, μέχρι το 2020 η περίοδος της υγιούς ζωής κατά δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι θα ζουν ανεξάρτητες και υγιείς ζωές σε προχωρημένη ηλικία, θα, μπορέσει να είναι, θα μπορέσουν να είναι πιο ολοκληρωμένα τα συστήματα ε, παροχής ιατρικής ε, φροντίδας και υπηρεσιών. Η έμφαση στην καινοτομία θα αποτελέσει ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας της. Η χρήση, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η καινοτομία θα αποτελέσει εξαιρετικό εργαλείο για να αντιμετωπιστούν δυσκολίες της γυράσκουσας κοινωνίας μας. Θα πρέπει η εταιρική αυτή σχέση να καλύψει κάποιους τομείς. Και η έρευνα σε αυτό προσκάλεσε πάνω από ε, πέντε συνεισφορές. Η διαθεσιμότητα του συστήματος υγείας είναι βασική, δεδομένου ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια γυράσκουσα Ευρώπη με περιορισμένους δημοσιονομικούς πόρους. Για να υπάρξει μια χρηματοοικονομική βιωσιμότητα θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόθεση της υγείας και την πρόληψη των παθήσεων για να αυξηθεί ο αριθμός των ετών που θα είμαστε υγιείς. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο καλά τους διαθέσιμους πόρους ώστε η υγεία του πληθυσμού να, να βελτιωθεί χωρίς να αυξηθεί ο προπολογισμό της υγείας. Θα πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία που μας προσφέρει η Ευρώπη 2020 να εξασφαλίσουμε τους, ε, τους, τους όρους της ε, παγκοσμιότητας, της καλής υγείας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Ένα σημαντικό τρόπο να επιτευχθεί αυτό είναι να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να τονίσουν όλο και περισσότερο το θέμα τη υγεία στου περαιτέρω γύρου ε, μεταρρύθμιση. Η στήριξη του Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά είναι ευπρόσδεκτη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είμαι πεπισμένος ότι παίζεται σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση ε, ε, του να στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των καταναλωτών η εργασία των θεσμικών μας οργάνων. Γι' αυτό θέλω να εξασφαλίσω ότι οι συντονισμένες προσπάθειές μας θα προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες μας. Και τώρα προσβλέπω στις απόψεις και τις ερωτήσεις σας σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλο χειροκρότημα από τα μέλη της Επιτροπής. Δεν συμβαίνει πάντα όταν μιλάει Επίτροπος εδώ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Ντάλι για το ευρύ φάσμα θεμάτων που καλύψατε και ορισμένα από αυτά είναι δύσκολα όπως γνωρίζουμε και άλλα πιο συνενετικά και πιο εύκολα. Ε, τώρα, όσα θέματα αναφέρετε, άλλους τόσους έχουμε μιλητές, 23 επικίνδυνη επιστολή πριν τις 4. Θα πρέπει να είμαι ε, πάρα πολύ αυστηρός, δύο λεπτά και τίποτα παραπάνω. Ε, να κάνετε ερωτήσεις και όχι ε, σχόλια. Ο Πέτερ Λίζε, πρώτος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε, κύριε Ντάλι για την παρουσίαση και για τη συνεργασία που έχουμε στο ένα, ένα χρόνο και κάτι. Στην ακρόασή σας ε, είπατε ότι θα λάβετε πρωτοβουλίες με θέμα τις ανεξάρτητες οργανώσεις ασθενών. Δηλαδή πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι πραγματικά ανεξάρτητες αυτές οι οργανώσεις από μεμονωμένες φαρμακευτικές εταιρείες και πώς μπορούμε να τους ε, βοηθήσουμε και πώς μπορείτε εσείς να εργαστείτε καλύτερα προς όφελος των ασθενών. Ξέρω ότι έχετε κάνει προσπάθειες ε, σε αυτό το τομέα, αλλά το επόμενο διάστημα ποια συγκεκριμένα βήματα μπορούμε να περιμένουμε, παρακαλώ. Ένα δεύτερο θέμα που απασχολεί πολλούς εδώ είναι τι γίνεται τώρα με την κλωνοποίηση και τα νέα τρόφιμα. Όλοι λυπούμαστε που να βάγισε η συνδιαλλαγή, ο καθένα έχει τη δική του ανάλυση για το τι πταίει ή τι πταίει. Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός και παραμένει ότι πολλά πράγματα ήταν ε, συνενετικά. Βέβαια υπάρχει και ένα ε, μεγάλο δηλαδή πεδίο που θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε εύκολα για τη συνέχεια και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Οκτωβρίου εξακολουθεί να ισχύει. Γιατί δεν είναι μόνο υποχρεώσει απέναντι σε άλλα θεσμικά όργανα, αλλά και απέναντι στην κοινή γνώμη και στου τομεί της οικονομίας που ενέχονται εκεί. Πώς θα προχωρήσουμε. Δύο προτάσεις τώρα θα φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν ε, σκέψεις ίσως και κάποιο χρονοδιάγραμμα ή τι μπορούμε αυτό που μας ένωσε να το ξαναφέρουμε. Ευχαριστώ. Πρόταση. 1,5 λεπτό το δίλεπτο. Η Λίντα Μακέβαν. Okay. Yes, I was going to ask about cloning. Ναι, εγώ θα ρωτούσα για την κλωνοποίηση. Τι γίνεται λοιπόν με την κλωνοποίηση. Ε, ακούγονται διάφορες φήμες ότι θα γίνει κάτι με την οδηγία για τα καλλιτικά. Πολλοί πίεση από τις εταιρείε προσπαθούν να αλλάξουν την προθεσμία. Μπορείτε να μας πείτε τι σκοπεύει να κάνει ή τι δεν σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν. Και τέλος, για το πακέτο για το κρέα. Είχαμε μία πρόταση πριν τα Χριστούγεννα που κατέστησε σαφές ότι θέλουμε να μείνει η, το, η επιθεώρηση για το κόκκινο κρέα, Θέλουμε ανεξάρτητες, ε, ανεξάρτητους ελέγχους και όχι εταιρείε. Η κυρία Ρης, ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά τα θέματα, έχουμε λίγο χρόνο. Θέλω να... Ε, σε, δεν ξέρω αν όλοι, τους, ε, αν όλοι οι συνάδελφοι πνίγονται, όπως και εγώ στο γραφείο μου, από τις διάφορες εγκλήσεις όσον αφορά τα παραδοσιακά φάρμακα επί τη βάση φυτών χιλιάδες mail, αιτήσεις, ε, αναφορές και φυσικά όταν κανείς το ψάξει λίγο το θέμα διαπιστώνει πως κάποιος ε, που θέλει να τα προωθήσει βρίσκεται σε αυτό, το, στη βάση αυτής της, αυτών των αναφορών. Πρόκειται για την οδηγία που αφορά τα παραδοσιακά φάρμακα με βάση φυτά και που σύμφωνα με αυτές τις αναφορές η οδηγία εμποδίζει την πρόσβαση σε εκατομμύρια λέει, καταναλωτές σε αυτά τα παραδοσιακά φάρμακα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω με ποιο τρόπο η ε, Κομισιόν θα απαντήσει σε αυτή θεμητή, το θεμητή ε, ανησυχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι αλήθεια ότι πνίγονται στην περιπλοκότητα των ευρωπαϊκών κανόνων. Πώς λοιπόν τους απαντάτε, πώς ε, διαρθώνεται η επικοινωνία με την Κομισιόν, γιατί εγώ διάβασα τις απαντήσεις της Κομισιόν και εγώ εδώ μιλώ για τους πολίτες και όχι για τις επιχειρήσεις του τομέα. Είναι λίγο ε, αλαμπουρνέζικα αυτά που λέτε που τους απαντάτε. Πολλοί πολίτες χρειάζονται αυτού του είδους τα φάρμακα. Ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση για την ε, βιοπικιλότητα λέει η κυρία Γκέρλινγκ. Στην ε, δική μου επικράτεια έχουμε διάφορα καλά προγράμματα με το Life ε, Plus και θέλαμε να είπατε ότι μπορεί να εισαχθούν διάφορα καινοτόμα δημοσιονομικά μέσα. Τι είδους μέσα θα είναι αυτά ε, και πώς πιστεύετε πως αυτά θα, θα προσελκύσουν χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα για τη βιοπικιλότητα. Ισα του χάσει. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω ποιο είναι το πρόγραμμα του Επιτρόπου σε σχέση με τα νέα τρόφιμα και την κλωνοποίηση των ζώων. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας και κατάλαβα καλά ότι με την υφιστάμενη νομοθεσία πρέπει να υπάρχει έγκριση πριν την αγορά, πριν να μπορέσει να απολυθεί οτιδήποτε που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα στους καταναλωτές. Κάτι άλλο αφορά την αρκοληψία και την ε, εμβολιασμό για την ε, ε, γρήπη των χείρων. Υπάρχουν τουλάχιστον τρει χώρε όπου έχουν με δει να αυξάνονται τα περιστατικά ναρκοληψία σε παιδιά αφού ε, έγινε ο εμβολιασμό για την γρήπη των χείρων. Εμένα με εντυπωσιάζει ο ρόλος της ε, Κομισιόν, διότι η Κομισιόν θα έπρεπε να είναι ο διαχειριστή του κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων δίνει μια γνωμοδότηση για την αδειοδότηση, αλλά η Κομισιόν λαμβάνει την απόφαση για τις αδειοδοτήσεις. Μέχρι στιγμής η Κομισιόν δεν έχει λάβει νέα απόφαση για τον εμβολιασμό για αυτή την πανδημία, αν και για παράδειγμα στη Φιλανδία σταμάτησε αμέσως ο εμβολιασμός όταν παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός περιστατικών αρκοληψίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ματίας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που μας παρουσίασε τους προσανατολισμούς για το 2012. Ορισμένα ερωτήματα που ήθελα να υποβάλω ήδη υποβλήθησαν και δεν θέλω να τα επαναλάβω. Γι' αυτό επιτρέψτε μου κύριε Επίτροπε να στραφώ λίγο στα λεπτομέρειες, σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες βασικά. Εσείς μας παρουσιάσατε τις διαδικασίες συναπόφασης στο, που, στη χρονιά που μας πέρασε τις προτάσεις οδηγιών που ήταν πιο σημαντικές και ήθελα να ρωτήσω ποια είναι, ποιος είναι ο στόχος ε, της Κομισιόν όσον αφορά κάποια θέματα που δεν είναι θέματα στην αλλά που ξεκινάνε από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου μέσω ψηφισμάτων, όπως για παράδειγμα το ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του Αλσχάιμερ και άλλων ε, τύπων άνοιας. Ε, τι είδου συνέχεια θα δώσετε όσον αφορά την ε, εφαρμογή ορισμένων πρωτοβουλειών του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Μας παρουσιάσατε ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον για το 2012 και τόσο το καλύτερο γιατί θα έχουμε θέματα πολύ σημαντικά. Εγώ θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση μετά από την υπόθεση Μεντιατόρ στη Γαλλία και για, για τα δυσδοκιμές αντοχής σε σχέση με το Μεντιατόρ και την ενημέρωση των ε, ασθενών. Πρόσφατα κάνατε προτάσεις μετά από αυτά τα τεστ ανοχής, πέρα από την ε, εντατικοποίηση της εποπτείας των φαρμάκων, ε, μιλάτε για περισσότερη διαφάνεια, είπατε ότι θέλετε να ενισχύσετε την ευρωπαϊκή διαδικασία επίγουσας απόσυρσης φαρμάκων από την αγορά, αλλά πώς θέλετε να μεταφράσετε σε πράξη όλες αυτές τις προτάσεις, ποια είναι τα νομοθετικά μέσα που θα χρησιμοποιήσετε και τόσο να αφορά την ενημέρωση των ασθενών, που βρίσκεστε, οι προτάσεις ε, αναμένονταν για τον Μάιο έχουν ήδη αναβληθεί πολλές φορές. Θα ήταν λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε τι προτίθεστε να μας πείτε για το μέλλον, για, μάλλον σύντομα, και πότε θα δημοσιεύσετε αυτές τις προτάσεις σας. Ο κύριος Γιώργενσον, ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Ε, ξέρω ότι ασχολείστε ιδιαίτερα με την ευημερία των ζώων και αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον έναν οδικό χάρτη για την ευημερία των ζώων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε πολλές συγκεκριμένες προτάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, τίποτα δεν συμβαίνει, δεν κινείται τίποτα. Μήπω μπορείτε να μας πείτε τι μπορούμε να περιμένουμε. Θα υπάρξουν προτάσεις από πλευρά σας φέτος. Και για ένα συγκεκριμένο θέμα για τη μεταφορά των ζώων. Το 2005 ο Επίτροπος Κυπριανού είχε δηλώσει ότι θα επρότεινε νομοθεσία μέχρι το τέλος της θητείας του. Αργότερα η Επίτροπος Βασιλείου μας διαβεβαίωσε ότι και εκείνη θα μας έκανε προτάσεις. Κανένας όμως τελικά δεν έκανε τίποτα. Τώρα, ξέρω, θα μας πείτε, χρειάζονται περισσότερες μελέτες επιπτώσεων, περισσότερες εκθέσεις. Εάν δείτε όμω τι εκθέσει των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση αυτή τη νομοθεσία και την επιβολή τη, θα δείτε ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερε εκθέσει, αλλά νέα νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί μάλιστα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ο κύριο Γκερμπράντι. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ντάλη. Η ερώτησή μου αφορά αυτό που είπατε για τον νόμο για την υγεία των ζώων. Είπατε ότι θα φέρετε του χρόνου νέε ιδέε σχετικά και μιλάτε για την πρόληψη, ότι είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Και θα αναθεωρήσετε τα κτηνιατρικά φάρμακα και θέλετε να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα τέτοιων φαρμάκων. Ερωτώ. Το εξής, ότι έχουμε υπερβολική χρήση αντιβιωτικών στην κτηνιατρική. Το πρόβλημα αντίνεται γιατί ο κόσμος τελικά ε, αναπτύσσει αντοχή και αντίσταση στα αντιβιωτικά, γιατί χρησιμοποιούνται αυτά κατά κόρον και στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Θα κάνετε πιο αυστηρή ε, την νομοθεσία για τη χρήση των αντιβιωτικών στη γεωργία γέννη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυλακάκης, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε, κύριε Πίτροπρα. Είναι πολύ σωστή η χρονική αλληλουχία, γιατί και εγώ για τα αντιβιωτικά θέλω να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 400.000 ασθενείς οι οποίοι έχουν ε, αντοχή ε, σε πολλά αντιβιωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το πρόβλημα των αντιβιωτικών όχι μόνο στο τομέα της κτηνοτροφίας αλλά και στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και στα κράτη-μέλη αλλά και σε πολλά μη κράτη-μέλη. Υπάρχει έλλειψη στον τομέα της έρευνας για νέα αντιβιωτικά. Η κατάσταση επιδεινώνεται σταθερά χρόνο με το χρόνο. Το βλέπουμε να έρχεται το κακό και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να υπάρχει κάτι το εξαιρετικό. Μία φουκουσίμα σε ένα εξαιρετικά ανθεκτικό μικρόβιο, το οποίο μπορεί να μην μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα, αλλά είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Όσον αφορά το θέμα της επικουρικότητας, η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 168 άρθρο αναφέρει ότι τα μεγάλα, τα σοβαρά διαμεθοριακά προβλήματα υγείας μπορούν και πρέπει να αφορούν την Ευρώπη. Τι έχετε να προτείνετε σχετικά. Ευχαριστώ κυρία Ροτμπέρεντ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ τον Επίτροπο στα αγγλικά. Οι τελευταίες μας ε, συναντήσεις κάπως επισκιάστηκαν από διάφορα γεγονότα. Ελπίζουμε τώρα να προχωρήσουμε με νέα πνοή. Και θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε τώρα. Θα φέρετε μια νέα νομοθετική πρόταση για το novel food, για τα νέα τρόφιμα, μαζί με την κλωνοποίηση, χωριστά. Τι θα την κάνετε την κλωνοποίηση. Ε, αν θα φέρετε ειδική πρόταση, αν όχι γιατί και ποιες δυνατότητες ιχνηλασιμότητας ε, έχετε ήδη προβλέψει για το σπέρμα, για τα έμβρια των ζώων κτλ. Τουλάχιστον την επισήμεση όλων αυτών των θεμάτων που ε, θα μπορούσαν να επανέλθουν όπως έγινε με το Novel Food. Επειδή μιλάω πάρα πολύ γρήγορα στα αγγλικά και δεν είναι η μητρική μου, έχω λίγο χρόνο και επανέρχομαι στην νομοθεσία για τα καλλιντικά, όπου η Λίντα Μακάβαν είχε την καλοσύνη να τα αναφέρει. Υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Η νομοθεσία και τελευταία τροποποίηση είναι και δεσμευτική. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι θα τηρηθούν οι προθεσμίες και δεν έχουμε διάφορα παραθυράκια. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορη και μέσα στο χρόνο σου. Επόμενη, κυρία Λεπάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους, κύριο Συντάγμαρ, για το θέμα της κλωνοποίησης. Είναι κατεπήγον. Έχει Έχουν προκληθεί ανησυχίε στην Ευρώπη από τους καταναλωτές για να δούμε αν τρώμε κλωνοποιημένο κρέας ή όχι. Πράγματι, είναι κατεπηγόντως ε, να, ανάγκη να δοθεί μια διευκρίνηση για τους γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς ως συγγήτρια κύριε Επίτροπε, σαφώ είμαι στη διάθεσή σα για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένου ότι πλέον υπάρχει η έκθεση τη Επιτροπής Περιβάλλοντος πια. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση και πάλι της ΕΦΣΑ, αλλά μια συμπληρωματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως συμβαίνει και με τα ζυζανιοκτώνα. Και φτάνουμε στο επόμενο θέμα που βρισκόμαστε με τις κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία όπως και για το περιβάλλον όσον αφορά για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Σας συγχαίρω για τη στάση σας, αλλά ε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, τι θα κάνουμε με την αρχή της ε, συγκριτικής αξιολόγησης ασφαλείας και αν είστε πάντοτε διατεθειμένος να αναθεωρήσετε το θέμα των εμπειρογνωμόνων για να αποφύγουμε την διαπλοκή στο πλαίσιο της επιστήμης ώστε να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους οργανισμούς, στον οργανισμό που χρειαζόμαστε, δηλαδή την ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ. Πρώτον, Συμφωνώ με τους συναδέλφους για τις νέες τροφές. Κλωνοποίηση των ζώων, των απογόνων του η χνηλασιμότητα, χρονοδιάγραμμα που έχετε για να κινηθείτε από αυτού δεδομένου του κατεπήγοντος χαρακτήρα. Δεύτερον, έχετε σκοπό να προχωρήσετε με την ευρωπαϊκή ε, συνταγογράφηση για φάρμακα. Τρίτον, όσον αφορά την υγεία των ζώων, τι χρονοδιάγραμμα έχετε θέσει. Σκοπεύετε να εισάγετε ένα μητρό ζώων συντροφιάς. Ευχαριστώ, Σφίμπτ. Η uh, Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε Νταλή, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θα ήθελα σύντομα να σας μιλήσω για το ψήφισμα Ε, για, όπου είχαμε μεν πλειοψηφία αλλά δεν είχαμε την απαραίτητη πλειοψηφία για να σταματήσουμε αυτήν την, ε, την διαμαρτυρία ε, σε σχέση με την DHA. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, είναι το θέμα γενικότερα όσον αφορά τους ισχυρισμούς των διαφόρων φαρμάκων. Θέλω να μας πείτε όμως ποια βήματα θα ακολουθήσετε ώστε να είστε βέβαιοι ότι ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα είναι υπέρ των παιδιών και των ε, γονιών τους εδώ στην Ευρώπη, διότι κάποιες φορές οι πόροι που χρησιμοποιούν οι ομάδες πίεσης είναι τεράστιοι και οι ΜΚΟ δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ώστε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να είναι προς το συμφέρον των παιδιών και όχι απαραίτητο των ε, κατασκευαστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. κύριο ε, κύριος Περέιο. Με κάλυψαν κάποιοι συνάδελφοι, οπότε σε εκμεταλλευτώ το λίγο χρόνο που έχω για να σας αναφέρω μια ανησυχία και μια ερώτηση. Επιλέγεται τώρα ο διευθυντής της υπηρεσίας για τα φάρμακα, όπως έγιναν και άλλοι διορισμοί. Και ανησυχώ γιατί βλέπω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ε, να έχουν θέσει υποψηφιότητες ή υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν μπορούμε για λόγους διαφάνειας να βάλουμε κάποιους κανόνες για να μην έχουμε αυτό το είδος ε, της διαπλοκής, γιατί άμα βάζεις ένα διοικητικό συμβούλιο να επιλέγει διευθυντή, θα επιλέξει από τους δικούς του. Είναι άλλοι έξι να του ομαδοποιήσουμε και να απαντήσετε εσεί συνολικά, συνθετικά στο τέλο. Μάλιστα, λέει ο Επίτροπο. Κριστιαν Μποζόη. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, να συγχαρώ τον Επίτροπο Ντάλι για την αφοσίωσή του και την δραστηριότητα που δείχνει όχι μόνο στον τομέα της δημόσια υγεία, αλλά και τη προστασία των καταναλωτών. Δύο ερωτήσει. Και μια τρίτη που όμως καλύφθηκε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ήθελα για την πρωτοβουλία σας για τις μεταδοτικές ασθένειες. Είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τα διαμεθοριακά θέματα υγείας αποτελεσματικά. Ξέρω ότι το έχετε στο πρόγραμμά σας. Μήπως μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεύτερον, θέλω να σας συγχαρώ που αποφασίσατε να αναθεωρήσετε την οδηγία για τις κλινικές δοκιμές. Δεδομένου, η φυστάμενη νομοθεσία μάλλον εμποδίζει την καινοτομία παρά τη στηρίζει. Και αν σε κάποια κράτη-μέλη οι κλινικές δοκιμές πάνε καλά, το βασικό πρόβλημα αφορά τις ε, πολυεθνικές, τα πολυεθνικό σκέλος γιατί η διαδικασία έγκρισης και αξιολόγησης έχει πολλά γραφειοκρατικά βάρη. Τι ακριβώς θέλετε να βελτιώσετε ε, σε αυτό το τομέα και δεδομένου ότι κάναμε την, ε, το σχέδιο γνωμοδότηση από την πλευρά της Επιτροπής συμφωνώ και εγώ με την κυρία Γκροστέτ. Θέλω να μας πείτε πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα της οδηγίας η οποία δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Ευχαριστώ. Βέσλετ. Νομίζω ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται η πώληση ψαριών με υψηλά επίπεδα διοξίνης. Όμως η και Φιλανδία έχουν εξαίρεση. Και εκεί είναι επίσης δυνατόν να πουληθούν ψάρια από την Βαλτική που, όπου η συγκέντρωση διοξίνης είναι υψηλή. Υπάρχει μια τάση επέκτασης και φαίνεται ότι η Κομισιόν θα δεχτεί αυτή την πρόταση. Υπάρχουν όμως δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να ενημερωθούν οι καταναλωτές ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να καταναλώσουν υπερβολική ποσότητα διοξίνης. Και πρέπει να γνωρίζουμε πόσο δηλητήριο πόσο δηλητηριώδης μάλλον είναι η διοξίνη. Παρά τα αυτά, χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες έμβρια είναι εκτεθειμένα στη διοξίνη. Και γνωρίζουμε ότι παρά την απαγόρευση αυτά τα ψάρια εξάγονται και εκατοντάδες κιλά ε, αυτών των ψαριών που περιέχουν διοξίνη πήγαν στη Γαλλία. Θέλετε να χορηγήσετε αυτή την εξαίρεση και στην Σουηδία, θα το κάνετε. Ο Καρλ Σλούτερ και Ιώσ, παρακαλώ. Uh, να σας ρωτήσω καταρχήν, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις, παραθυράκια, τίποτα όσον αφορά τις συστοιχίες ε, κλοβών, και ότι θα επιβληθούν ποινέ σε όσους δεν το εφαρμόνουν το, ίδιο για τα καλλιτικά. Καμία παράταση, καμία, κάνα παραθυράκι, καμία εξαίρεση. 2013 να είναι η τελική διορία. Μπορείτε να μου το εξασφαλίσετε αυτό και έπειτα για τα τρόφιμα και για την ραδιενέργεια. Η Ευρατόμ το χρησιμοποιεί. Ε, το χάσει το ραδιοενεργό υλικό της η, η πυρηνική βιομηχανία. Η ΣΑΝΚΟ θα πρέπει να ασχοληθεί. Θέλετε να, να αλλάξετε την νομική βάση για αυτή τη δικασία και έπειτα για την μεταφορά ζώων. Ξέρετε ότι τη θέση δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Τουλάχιστον όλα τα 27 κράτη ε, παραβιάζουν την σχετική νομοθεσία, ίσως με την εξαίρεση της Μάλτας. Όλοι παραβιάζουν αυτή τη νομοθεσία. Παρακαλώ να εξασφαλίσετε την πλήρη εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν συμφωνούσε απολύτω ο γιο σου. Ε, τι ήταν το σχόλιο, μου ξέφυγε. Πάντω αυτό το κατάλαβε. Ο Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, η στρατηγική για την υγεία 2012-2013 είναι καλή και μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί καλά. Και τώρα έρχεστε να μας φέρετε μια δεύτερη ανακοίνωση κάποια στιγμή για το δεύτερο στάδιο. Μπορείτε να μας πείτε τι θα κάνετε με το, νομοσχέδιο, το νόμο για την υγεία των ζώων. Κάτι άλλο που είναι ακαθόδες είναι το κόστος για τους επίσημους κρατικούς ελέγχους. Από χώρα σε χώρα αυτό διαφέρει. Υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού και ε, θα πρέπει πολύ γρήγορα να βρούμε κάποια ρύθμιση έτσι ώστε να αρθούν αυτές οι ανομαλίες. Και τώρα η κρεοσκοπική έλεγχη και πάλι η κρατική και η επίσημη. Υπάρχουν ε, ζωνώσει ε, που δεν αναγνωρίζονται πάντα, δεν εντοπίζονται πάντα σε ελέγχους, χρειάζονται νέες μέθοδοι. Πώς θα τις προωθήσετε αυτές. Επίσης, ε, ακούσαμε ότι είναι δύσκολο κάπου να ε, αποδοθούν οι ευθύνε για την αντίσταση στα αντιβιωτικά. Άλλοι ρίχνουν την ευθύνη στα ζώα, άλλοι στον άνθρωπο. Θα πρέπει να γίνουν και εδώ νέε έρευνε και να το προωθήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην παίρνουμε λάθο αποφάσει ε, στο νομοθετικό πεδίο. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα των διοξινών. Είπατε πρόσφατα ότι θέλετε να δείτε ε, πώς θα χωρίσετε τις μεθόδους παραγωγής και ε, το, αυτό το έχετε προχωρήσει και πού έχετε φτάσει. Ευχαριστώ. Ο Κρήτον Αρσένης, παρακαλώ. Thank you very much. a lot of scandals in the EFSA. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς ήδη στην αίθουσα είπατε ότι πρέπει να ανεξηγηθεί η ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε άλλο ένα ε, σκάνδαλο στην EMA που, θύχθη, που, που, αφορούσε έναν πρώην ε, ο διευθυντή ο οποίος μετακινήθηκε στην ε, γεωργική βιομηχανία. Φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα λοιπόν στις αρχές που αποφασίζουν για την υγεία μας και για κρίσιμες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Τι θα κάνετε για αυτά όλα. Πώς... Ε, και πότε θα αρχίσουν να δουλεύουν σωστά αυτές οι υπηρεσίες, αυτοί οι οργανισμοί. Και έπειτα, για την Ιαπωνία. 12 από τις 27 νομαρχίες αναγκάζονται να ελέγξουν τα τρόφιμά τους πριν τα στείλουν στην Ευρώπη. Δεδομένη της κλίμακας αυτού του ατυχήματος, θα ζητήσετε αυτές οι δοκιμές να γίνονται και για τα προϊόντα που προέρχονται από άλλες νομαρχίες της Ιαπωνίας. Ευχαριστώ. Last ο Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταρχήν και εγώ ήθελα να αναφέρω το πρόβλημα των ασθενειών που αντιστέκονται στα φάρμακα. Το Νομίζω πως θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών. Δεύτερον, για το καπνό. Σωστά υπογραμμίσατε την τοξικότητα που συνδέεται όμως και στην, ε, στο, στον τρόπο ε, της... Ε, τη, της χρήσης του καπνού, κυρίως δηλαδή μέσω της αναπνοής, της εισπνοής, με συγχωρείτε. τι θα κάνετε όμως και για άλλα είδο χρήσης του καπνού, όπως ας πούμε τον καπνό που χρησιμοποιείται υπογλώσια. Τώρα, για το σύστημα των ανοσοποιητικών, τι άλλο προετοιμάζει η Κομισιόν σχετικά με τον καπνό. Ρώτησε ο Βιτόριο Πρόντι. Τι είναι όταν έχει κάποιο καπνό υπογλώσιο. Γιατί μα στέλνουν οι Σουηδοί επιστολέ. Ξέρετε ότι οι Σουηδοί σνιφάρουν καπνό και φωνάζουν όταν θέλουμε να το εντάξουμε στα τσιγάρα, όπω το κάπνισμα. Το 2006 αποφασίσαμε με ένα νόμο για τι βιταμίνε και τα μεταλλικά άλατα ε, και τα ιχνοστοιχεία ε, στα τρόφιμα και μέχρι το 2009 επρόκειτο να ορίσετε τις ανώτατες τιμές. Τώρα είμαστε Απρίλιο του 2011. Να περιμένουμε τίποτα από εκεί υπάρχουν προβλήματα. Ορίστε, έχετε ένα ολόκληρο φάσμα, ένα ποτ πουρί ερωτήσεων. Καλή τύχη στις απαντήσεις, παρακαλώ. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον και για σας να ακούσετε όλο αυτό το φάσμα των ανησυχιών και των μελημάτων των μέλων μας. Ε, παρακαλώ, απαντήστε. Πράγματι ήταν πολύ ενδιαφέρον με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα όλες τις απόψεις. Αυτού του είδους η συζήτηση πραγματικά μας βοηθάει για να επιλέξουμε κατευθύνσεις και προτεραιότητες. Πραγματικά μπορούμε να αισθανθούμε τη σκέψη του Κοινοβουλίου και ποιες είναι οι προτεραιότητες που τον, το ενδιαφέρουν όπως επίσης και τα προγράμματα στα οποία θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Θέλω επίσης να σας συγχαρώ για την πειθαρχία που δείξατε. Όλοι μιλήσατε εντός των ορίων του χρόνου που σας δόθηκε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σχολιάσω τα θέματα που τέθηκαν. Πρώτον, για τις οργανώσεις των ε, ασθενών και τους ε, προπολογισμού και την ανεξαρτησία. Πώς θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο, να εξασφαλίσουμε ανεξαρτησία από των οργανώσεων των ασθενών όπως και των οργανώσεων καταναλωτών και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε τους αυστηρούς περιορισμούς για... στο δημοσιονομικό επίπεδο που μας επιβάλλονται. Πράγματι, πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα. Όπως σας έχω υποσχεθεί κατά την ακρόαση μου και όπως μου υπενθύμησε και ο Πίτερ, υποσχέθηκα ότι θα προσπαθήσω να βρω νέους τρόπους για να δούμε πώς μπορούν να ρεύσουν πόροι σε, αυτούς τους, σε αυτές τις οργανώσεις ασθενών χωρίς βεβαίως να υπονομεύσουμε την εξαρτησία τους. Το μελετήσαμε. Υπάρχουν φυσικά κάποια ζητήματα για τους κανονισμούς, τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς που ισχύουν και πρέπει να τα μελετήσουμε και αυτά. Δεν είναι εύκολο. Αν θέλουμε να μην υπάρχουν εμπορικές επιδοτήσεις στους οργανισμούς αυτούς, θα πρέπει να αυξήσουμε τις δημοσιονομικές ενισχύσεις, πράγμα που δεν φαίνεται εύκολο. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κάποιο είδος ταμείου, ίσως και ε, χρηματοδοτούμενο από τον ιδιωτικό τομέα, όπου όμως θα υπάρχει ένα φίλτρο μεταξύ των δωρητών και των ε, αποδεκτών. Να δούμε δηλαδή πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το δύσκολο θέμα. Ένα άλλο θέμα βεβαίως είναι οι νέες τροφές και η κλωνοποίηση. Σχετικά πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι το κατεπήγον του πράγματος. Η αξιοπιστία μας ως θεσμικό όργανο, ως Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα κινηθούμε. Χάσαμε ή εν πάση περιπτώσει αναστήλαμε την αναθεώρηση της οδηγίας για τις νέες τροφές, τα novel foods. Αυτό ήταν κάτι το πολύ καλό για την Ευρώπη. Πιστεύω ότι δεν καταφέραμε και να αυξήσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για το, την κλωνοποίηση των ζώων. Τι θα κάνουμε. Θέλω να υποβάλω το ταχύτερο δυνατόν ένα νέο νομοθετικό πακέτο που να αφορά την οδηγία των νέων τροφών και να αρχίσω να εργάζομαι, όπως είχα προ... υποσχεθεί και στην ε, διαβούλευση, να δουλεύω και να υποβάλω μια νομοθετική πρόταση εντός συγκεκριμένου διαστήματος που το έχουμε συζητήσει στην συνδιαλλαγή για το θέμα της κλωνοποίησης. Όμως, θέλω να προχωρήσω μαζί με σας. Ήδη έχω μιλήσει στην Επιτροπή Γεωργία σήμερα το πρωί και είπα ακριβώ το ίδιο. Θέλω να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσω ότι θα κινηθούμε προς μία κατεύθυνση και να εξασφαλίσουμε ταχεία επίλυση του ζητήματος. Δεν θέλω να υποψιάζεται κανένας ότι προσπαθούμε να παρακάψουμε το θέμα της κλωνοποίησης προχωρώντας στο θέμα των νέων τροφών. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Η ιδέα είναι ότι υπάρχει οδηγία των νέων τροφών, έχει συμφωνηθεί, κρίμα που δεν εφαρμόζεται. Ας εφαρμόσουμε μια ανάλυση, ας δεσμευτούμε και εγώ μπορώ να δεσμευτώ για το πώς θα προχωρήσουμε στο θέμα της κλωνοποίησης και είμαι διατεθειμένος να προχωρήσω. Ας το συζητήσουμε αυτό για να δούμε πού θα πάμε. Θέλω όμως αυτό να έχει επιληθεί πριν το τέλος του χρόνου, το ταχύτερο δυνατόν. Θέλω να κινηθώ γρήγορα επ' αυτού, γιατί αισθάνομαι ότι το χρωστάμε στους πολίτες μας τώρα οδηγία για τα καλλιντικά, χρονοδιαγράμματα, ε, τα χέρια και τα κλουβιά κλπ. Πιστεύω ότι πρέπει να το πιέσουμε. Υπάρχουν ε, οι μεταβατικές περίοδοι για να τηρούνται. Αυτό ισχύει για κάθε νομοθετικό κείμενο. Αν απλώς αναβάλουμε τις προθεσμίες, τότε η νομοθεσία μας δεν είναι αξιόπιστη. Αυτό ισχύει και στην νομοθεσία που καλύπτει για τα βοτανά τα ιατρικά βότανα. Εδώ είχαμε μια μεταβατική περίοδο 7 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας όλη η παραγωγή τέτοιων φαρμάκων με βότανα θα έπρεπε να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους. Το σύστημα της καταχώρησης, η διαδικασία καταχώρησης, ελαφρύνθηκε, διευκολύνθηκε, έγινε πιο φιλική προς τον χρήστη για χάρη τους. Η νομοθεσία, ας πούμε, σχετικά θεωρούσε ότι τα παραδοσιακά φάρμακα, αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί για πάνω από 30 χρόνια, θα μπορούσαν να καταχωρηθούν χωρίς να γίνουν ε, ιδιαίτερες αξιολογήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι και πάλι πάρα πολλοί ε, παραγωγοί τα τελευταία χρόνια, την 11η ώρα είπαν ότι δεν καταχώρησαν, δεν έκαναν τίποτα και ζήτησαν και άρχισαν να πιέζουν για μια παράταση της προθεσμίας, που δεν γίνεται. Έχουμε προχωρήσει γιατί έληξε η προθεσμία την 1η Απριλίου και αυτό είναι σωστό. Όσον αφορά τώρα τον τομέα των καλλιντικών, θα κάνουμε αυτό που προβλέπει η νομοθεσία. Η νομοθεσία προβλέπει ότι ήδη υπάρχει απαγόρευση δοκιμών, όπως γνωρίζετε έχει τεθεί ενισχύ, θα υπάρξει απαγόρευση εμπορίας, σε λίγους μήνες θα έλεγα, αλλά η Κομισιόν από την νομοθεσία πρέπει να αναφέρει για την κατάσταση των διαδικασιών δοκιμών. Πρέπει να πει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά τα, τις εναλλακτικές δυνατότητες. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Την έκθεση αυτή συντάσσουμε όπως ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία. Φυσικά, αυτό θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για να εκτιμήσουν την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τα κλουβιά, δύο φορές έχω επιμείνει στο Συμβούλιο. Δεν θα παρατείνω την προθεσμία, είπα. Όμως πρέπει να σας πω τι με ανησυχεί. Έχω ζητήσει από το Συμβούλιο να με ενημερώσει για, για το πώς πάμε όσον αφορά τη συμμόρφωση με αυτόν τον κανονισμό. Ήδη το έχω κάνει αυτό δύο φορές φέτος. Και μέχρι στιγμής υπάρχουν οκτώ χώρες που δεν μας έχουν ακόμα ενημερώσει για την συμμόρφωση με την νομοθεσία αυτή στην περιοχή τους. Στη Επιτροπή Γεωργίας αντιλαμβάνεστε ότι με βομβάρδισαν με ρωτήσεις για εναλλακτικά σχέδια Β, Γ, Δ κτλ. Όμως, όποιο σχέδιο και αν επιλέξω θα πρέπει να στηριχθώ σε στοιχεία, στην πραγματικότητα που, που υπάρχει στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να έχουμε 85 εκατομμύρια αυγά την ημέρα που να μην συμμορφώνονται με τον κανονισμό. 85 εκατομμύρια αυγά την ημέρα έχουν, που έχουν αγορά, καταναλώνονται, παράγονται από όρνηθες που τρώνε ζωοτροφές, άρα οι επιπτώσεις της οποιασδήποτε απόφασης μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Από την άλλη όμως πλευρά πρέπει να υπάρχει και κάποια βασική αντίληψη. Δηλαδή οι χώρες και οι παραγωγοί που συμμορφώθηκαν με τον κανονισμό δεν θα πρέπει να υποστούν διάκριση με αθέμητο ανταγωνισμό από αυτού οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κάνω είναι το εξή. Προσπαθώ να συγκεντρώσω και τι τελευταίε πληροφορίε ώστε να έχω την εικόνα της κατάστασης και να δω τις επιπτώσεις των ε, αποφάσεων που θα λάβουμε και θα επιστρέψω και πάλι σε εσά με προτάσεις για το τι θα πρέπει να κάνουμε. Για την αρκοληψία. Προς το παρόν, και αφού ενημερωθούμε για τα βρήματα αυτά, κυρίως από τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Νομίζω ότι και στη Γαλλία έχουν εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις. Ζητήσαμε από το ECDC που εργάζεται αυτή τη στιγμή για να κάνει μια αξιολόγηση κινδύνου σχετικά. Επίσης η ΕΜΑ ε, μελετά το θέμα. Έχουμε δύο λοιπόν αυτούς, αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα και περιμένουμε ενημέρωση από αυτούς. Το mediator είναι πρόβλημα. Πρόβλημα των εθνικών αρμοδίων αρχών έγκρισης φαρμάκων. Είναι μια υπόθεση την οποία παρακολούθησα το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών είχαμε συζήτηση με τον Γάλλο Υπουργό που παρουσίασε την κατάσταση στη Γαλλία προς το Συμβούλιο. Όταν άκουσα για το Μεντιατόρ έδωσα οδηγίες στις υπηρεσίες μου να κάνουν ένα τεστ αντοχής της νέας ε, νομοθεσίας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και ρώτησα αν ίσχυε αυτή η νέα νομοθεσία θα είχαμε την υπόθεση με διέτορ. Αναλύσαμε λοιπόν την κατάσταση και διαπιστώσαμε τρία θέματα που πρέπει να τα διορθώσουμε. Τρία ζητήματα είναι η νέα νομοθεσία που έχουμε μόλις ψηφίσει, δεν έχει καν τεθεί ενισχύει και παρά τα αυτά ήδη χρειάζονται να διορθωθούν τρία ζητήματα. Πρώτον, να φροντίσουμε πάντα να να υπάρχει ευρωπαϊκή διαδικασία σε περίπτωση εθνικής απόσυρσης. Δηλαδή να επιμένουμε ότι αυτό θα ισχύει σε κάθε περίπτωση. Δεύτερον, υποχρέωση του κλάδου να δηλώνει τους λόγους της απόσυρσης. Το πρόβλημα του Mediator ήταν ότι αποσύρθηκε εθελοντικά από πολλές χώρες, εθελοντικά, από την, επιχει... από την εταιρεία και η οποία επικεντρώθηκε κυρίως στη Γαλλία. Αυτό που ζητάμε η νομοθεσία να προβλέπει την υποχρέωση από τον κλάδο να εξηγεί για ποιο λόγο αποσύρεται το φάρμακο όταν αποσύρεται εθελοντικά. Και τρίτον, η δημοσίευση καταλόγου φαρμάκων που υπόκεινται σε παρακολούθηση μετά την θέση τους σε εμπορία. Άρα θέλουμε, επαναλαμβάνω, δημοσίευση καταλόγου φαρμάκων που υπόκεινται σε παρακολούθηση μετά την θέση τους σε εμπορία. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε την ομοθεσία μας ακόμα περισσότερο και ελπίζω ότι η υπόθεση Mediator δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Όσον αφορά την ενημέρωση των ασθενών τώρα. Μπορούμε να πούμε ότι η πρόθεση, η πρόταση και η διαδικασία μας προς την Κομισιόν και ελπίζω να τηρηθεί η προθεσμία του Μαΐου για την ε, δημοσίευση, το θέμα της ενημέρωσης των ασθενών. Το Κοινοβούλιο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά από αυτό, πιστεύω και συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό με το Κοινοβούλιο. Θα δείτε ότι οι προτάσεις μας δεν θα είναι ταυτόσιμες, αλλά πάρα πολύ παρόμοιες με αυτές του Κοινοβουλίου. Για την ευζοία των ζώων θα υποβάλουμε προτάσεις φέτος για να ενισχυθεί το καθεστώς ευζοίας των ζώων και να περιλάβει τι μεταφορά. Η έκθεση ήδη έχει καθυστερήσει για κάποιους ένα διάστημα για να εξασφαλίσουμε ότι θα συγκεντρωθούν επαρκή δεδομένα και στοιχεία ώστε να γίνει μια συγκεκριμένη μελέτη την, η οποία έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη και που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμεινο του 2011 και όχι ένα όπως είπε κατά λάθο ο Επίτροπος. Αυτή είναι μια διαδικασία, μια εργασία η οποία είναι υπό ολοκλήρωση. Αντιβιωτικά. Έχουμε μια ειδική μονάδα με, σε συνεργασία με την ECDC και εκεί συμμετέχουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε για να διαπιστώσουμε τι πρέπει να κάνουμε ε, το καλύτερο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των μικροβίων. Αποτελεί για μας θέμα προτεραιότητας επίσης. Και θα αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική τον Νοέμβρη του 2011. Συμφωνώ μαζί σας. Χρειάζεται να αναβιώσει, να δοθεί μια νέα όθηση στην έρευνα στο χώρο αυτό. Πρέπει να έχουμε εναλλακτικές λύσεις στα αντιμικροβιακά φάρμακα που υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στη χρήση των αντιβιωτικών, κυρίως στη γεωργία. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί, ε, να αντιμετωπίσουμε την κατάχρηση αυτών των φαρμάκων στις ζωοτροφές κλπ. Πακέτο υγιεινής. Όπως είπα, θα γίνει αναθεώρηση αυτού του πακέτου με διαδικασία συναπόφασης. Η έκθεση της Κομισιόν το 2009 για την εφαρμογή του πακέτου υγιεινής ε, ε, επισημαίνει την γενική ικανοποίηση των αρμοδίων αρχών και των επιχειρηματιών τροφίμων. Δεν θα υπάρξει γενική αναδιατύπωση του πακέτου. Βασικός στόχος της αναθεώρησης που κάνουμε είναι η εναρμόνιση της εφαρμογής κάποιων ορισμών του κρέατος, να γίνουν τελικές διατάξεις μεταβατικών μέτρων. Έχει γίνει ε, αναθεώρηση της επιθεώρησης κρέατος κάποιων στοιχείων της και έχει απλουστευθεί η γενική διαδικασία της συνθήκης. Σε, ε, μάλλον, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης, βεβαίως θα πρέπει να μείνει η επιθεώρηση και ο έλεγχος του κρέατος στα ε, χέρια των δημοσίων αρχών. Εδώ συμφωνούμε. ρωτήσατε για τις πρωτοβουλίες ε, υγείας. Το συζητήσαμε σήμερα το απόγευμα αυτό με τις υπηρεσίες μου, το πώς θα προχωρήσουμε. Μελετάμε νομοθετική πρόταση που θα υποβληθεί πριν το τέλος του έτους. Σκοπός μας είναι να γίνει υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη ή θα προτείνουμε, εν πάση περιπτώσει, να γίνει υποχρεωτικό. Να έχουν τα κράτη-μέλη ένα σχέδιο ετοιμότητας. Γιατί μέχρι τώρα αυτό είναι εθελοντική υπόθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών. Επίσης, η Επιτροπή Ασφάλειας της Υγείας θα πρέπει να επισημοποιηθεί. Υπήρχε μια άτυπη ρύθμιση, μια άτιμη δομή τα τελευταία χρόνια και ό,τι χρειαζόταν να μάθουμε τα τελευταία δέκα χρόνια το μάθαμε. Τώρα λοιπόν πρέπει να επισημοποιήσουμε την Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας. Μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για απειλές στην υγεία, ο πιο αδύναμος ε, κρίκος είναι το άθροισμα του συνόλου. Ένας να είναι ο δύναμος κρίκος όλης της αλυσίδας, αυτός καθορίζει τη δύναμη, την αντοχή όλης της αλυσίδας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είμαστε σε επιφυλακή, να υπάρχει επιφυλακή από κοινού. Επίσης θα συμπεριλάβει η διαχείριση κινδύνων και άλλους κινδύνους για να υπάρχει συντονισμός σε ανταπόκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι θέμα να αναλάβει η ECDC αυτές τις αξιολογίες κινδύνου, αλλά το συντονισμό της δράσης και η αξιολόγηση του κινδύνου θα μείνει σε επίπεδο κράτους μέλους. Όμως πρέπει να αρχίσει ε, μια καλύτερη οργάνωση για όλα αυτά όσον αφορά την καταχώρηση, την καταγραφή των ζώων συντροφιάς. Δεν ε, σκεφτόμαστε να εισάγουμε ένα τέτοιο μητρό, αλλά πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει διαβατήριο ζώων συντροφιάς. Καλύπτεστε, πιστεύω, όσον αφορά το θέμα αυτό. Για τα γενετικά τροποποιημένα, για τις γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αντιλαμβάνουμε σήμερα το πρωί, ε, ε, ψηφίσατε την έκθεση κυρίας Λαπάζ, Φυσικά θα μελετήσω αυτά που αποφασίστηκαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω γενικά για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εμπλεκόμενοι να ε, ε, συμμετέχουν σωστά και να αρέσκονται στην διαδικασία αδειοδότησης που προτείνουμε. Τώρα, οι προτάσεις της ΕΦΣΑ πριν από μερικούς μήνες έχουν πια μπει στο τραπέζι για να συζητηθούν και να μεληθούν από όλους. Έχουμε ήδη οργανώσει ή έχουμε συμμετάσχει σε δύο πολύ καλά σεμινάρια επ' αυτού. Προσκλήθηκαν πολιτικοί, επιστήμονες. Έγινε εξαιρετική συζήτηση. Προγραμματίζουμε τέσσερα ακόμα ε, σεμινάρια για να ασχοληθούμε με θέματα της ανεξαρτησίας, για την παρακολούθηση, τη διαθεσιμότητα των ε, δεδομένων προς όλους, ο περιορισμός αυτού του θέματος εμπιστευτικότητας να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο για να είναι ανεξάρτητη η μελέτη των δεδομένων και να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να κλείσω με ένα σύστημα, όχι που όλοι, αυτό είναι δυνατόν, αλλά που θα το εμπιστεύεται η πλειοψηφία, ότι είναι σωστό δοκιμές κλπ. κλπ. Και από αυτού θέλω να πω κάτι για την ΕΦΣΑ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για σκάνδαλα. Το τι σκάνδαλο ε, δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν, αλλά δεν είναι πάντα σκάνδαλα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και πάλι. Είναι ανησυχητική η κατάσταση και το γεγονός αυτό του προηγούμενου διευθυντού και μας ενόχλησε και μας και μένα προσωπικά πάρα πολύ. Το λέω δημόσια. Με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό. Και συνεργάστηκα και με τις υπηρεσίες μου για να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος την έρευνα. Πρέπει όμως να καταλάβετε κι εσείς το εξής. Αυτοί οι οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί. Εγώ ως Επίτροπος δεν μπορώ να υποχρεώσω ένα διοικητικό συμβούλιο τέτοιου οργανισμού και μιλάω και για την ΕΦΣΑ και για την ΕΜΑ να πάρουν την ΑΒ θέση. Είναι ανεξάρτητοι οι οργανισμοί. Δεν μπορώ να τους υποχρεώσω να επιλέξουν ένα πρόσωπο και να τον διορίσουν διευθυντή ή εκτελεστικό διευθυντή για να διευθύνει τον οργανισμό. Δεν μπορώ εγώ να τους επιβάλλω ένα πρόσωπο η απόφαση θα πρέπει να είναι δική τους. Και πολλές αποφάσεις ελήφθησαν που ε, δεν με βρίσκουν απαραίτητο σύμφωνο σε επίπεδο management διοίκηση. Λοιπόν, όμω είναι ανεξάρτητη και καλό είναι που είναι ανεξάρτητη, δεν διαφωνώ. Από την άλλη, όμω, πιστεύω ότι χρειάζεται αναθεώρηση του τρόπου με το οποίο διοικούνται αυτοί οι οργανισμοί. Και μπορώ να σας πω εδώ και εγώ ότι έκανα κάποιες προτάσεις ήδη ε, στους συναδέλφους μου και συγκεκριμένα στον Επίτροπο κύριο Σεύκοβιτς που ε, ασχολείται και είναι αρμοδιότητά του αυτά τα θέματα για να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Αυτό που θέλω εγώ για να ε, αυξηθεί και η λογοδοσία τους αλλά και η ανεξαρτησία τους. Ελπίζω να προχωρήσουμε προς την κατάσταση αυτή και θα βελτιωθεί. Επίσης, με ρωτούν ποιο θα είναι ο νέο εκτελεστικό διευθυντή στον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Με είναι δική του υπόθεση να το αποφασίσουν. Είναι πολλοί υποψήφοι. Πέρασαν από μια διαδικασία επιλογή συνεντεύξεων. Θα γίνει ένα σύντομο κατάλογο και βάσει αυτού του καταλόγου θα επιλεγεί ο Διευθυντή. Θα, θα δούμε. Κανόνες πάντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να τηρούνται οι κανόνες. Αν τηρούν τους κανόνες, ακόμα και αν η απόφαση αυτή δεν μας αρέσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ε, Έπρεπε να σας το πω αυτό. Εγώ δεν μπορώ να βάλω βέτο σε απόφαση που παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΑ. Πιέζουμε λοιπόν προς μια κατεύθυνση για να αναθεωρήσουμε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται αυτοί οι οργανισμοί, agencies. Για τις κλινικές δοκιμές, τι θέλουμε να βελτιώσουμε. Πολλά νομίζω μπορούν να βελτιωθούν εκεί. Υπάρχει μια οδηγία, την έχουμε δει στην πράξη να λειτουργεί και επίσης έχουμε ζήσει και θετικά στοιχεία ασφάλεια των ασθενών και η ιδεοντολογία ε, των κλινικών δοκιμών ε, πάρα πολύ ε, βελτιώθηκαν και ενισχύθηκαν. Από την άλλη έχουμε και δυναμίες όμως στον χρόνο εφαρμογής και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναφορά ή γενικά η οργάνωση είναι πολύ δύσκολο να κάνουν κλινικές δοκιμές χωρίς να απευθυνθούν οι εφερόμενοι καμιά φορά σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείε. Και αυτά είναι και φαινόμενα που δεν θέλουμε να συμβαίνουν. Μπορούμε να ελαφρύνουμε, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες και αυτό θα έκανε μεγάλο καλό σε πολλού. Για τα πυρηνικά ε, σας είπα, ο πρόεδρος Μπαρόσο την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο είπε ότι θα αναθεωρήσουμε τις ανώτατες τιμές για ε, τι πυρηνικές, ε, δηλαδή ενεργές ουσίες Αυτό τώρα πώς θα γίνει. Τώρα έχουμε αυτό το ζήτημα των πυρηνικών. Έχουμε μια οργάνωση από το Τσέρνομπιλ. Υπήρχε αυτό το σχέδιο. Πρέπει να αναθεωρηθεί, πρέπει να αλλάξει νομική βάση. Ε, και αυτό το βλέπουμε και το συζητάμε. Πάντως, κάτι πρέπει να γίνει. Μια ε, εμπειρογνωμοσύνη, γνωμοσύνη πρώτα απ' όλα και μετά για την πυρηνική τεχνολογία γέννη και στη συνέχεια τον επιστημονικό αντίκτυπο, πώς αυτό έχει επιπτώσει στα τρόφιμα. Μας αφορά βεβαίως και μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων αυτών. Διοξίνες. Και πάλι πιστεύω και έστειλα και ένα μικρό σημείωμα. Αυτό το επεισόδιο στη Γερμανία με τις διοξίνες, εμένα με παρηγόρησε ότι λειτουργεί σωστά το σύστημα. δηλαδή ότι καμία νομοθεσία δεν μπορεί να ε, προβλέψει κάποια εγκληματική δραστηριότητα όταν προσπαθεί κάποιος να το παρακάμψει. Πάντως όταν συμβαίνει αυτό έχουμε συστήματα ε, ανείχνευσης που λειτουργούν και πραγματικά τους πιάνουμε. Είναι σημαντικό αυτό και μας ενθαρρύνει να ενισχύσουμε το σύστημα. Βεβαίως χρειάζονται κάποιες αλλαγές να γίνουν, το συζητήσαμε με τη γερμανική κυβέρνηση και στο Συμβούλιο και προχωρούμε προς την έναρξη της εφαρμογής των όσων πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, για τη, τους ισχυρισμούς για το DHA. Έχουμε ε, απόφαση του Κοινοβουλίου και αυτή θα πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και πάλι για τους άλλους ισχυρισμού υγείας. Το θέμα είναι, τι θέλουμε, να ενδιαφέρονται ε, ε, οι αποφάσεις μας για τους πολίτες ή για τις εταιρείες. Τι μας ενδιαφέρει περισσότερο, τα συμφέροντα των καταναλωτών βεβαίως. Για τους ισχυρισμούς αυτούς υγείας ε, έχει εγκριθεί ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό τους. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει ή θα μπορούσε να καταγορηθεί η ΕΦΣΑ ότι αγωνίζεται για τη βιομηχανία σε αυτή την περίπτωση. Δεν ισχύει αυτό. Η μεγαλύτερη αντίδραση ε, τη βλέπουμε από τη βιομηχανία που είναι έξαλλη όταν αρνείται η ΕΦΣΑ κάποιες ε, μορφές ισχυρισμών τους να τις εγκρίνει. Και πραγματικά πολεμούν σκληρά και αγωνίζονται, αλλά εμείς κρατάμε γερά, δεν ενδίδουμε. Γίνονται αυτές οι ισχυρισμοί, ας πούμε, με επιστημονική βάση. Και έχουμε εγκρίνει έναν από τους λίγους ε, ισχυρισμούς υγείας, ε, λίγη είναι για να κυκλοφορήσει ένα ε, προϊόν στην αγορά. Και δεν είναι επιπόλαια η έγκριση. Υπάρχει επιστημονική βάση που τεκμηριώνει την έγκριση αυτή. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτή την υπόθεση ή να αφαιρέσουμε αυτό τον ισχυρισμό. Για τις βιταμίνες Γιώ, ε, αυτό που ρωτήσατε εσείς για τις βιταμίνες, ναι, ναι, το κοιτάμε, το εξεργαζόμαστε αυτό. for Α, για τις διοξίνες των ψαριών της Βαλτικής. Η Σουηδική κυβέρνηση όντως μας το ζήτησε. Όταν πήγα στη Σουηδία, ήταν από τα θέματα που μας απασχόλησαν εκεί και μου το έθεσαν υπόψη. Ζήτησε λοιπόν παράταση η Σουηδία της εξαίρεσης και προβλέπεται ψηφοφορία στην Επιτροπή τον άλλο μήνα. Και όντως η Σουηδική κυβέρνηση μας ενημερώνει ότι έχουν ειδική πληροφόρηση και ε, πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παιδιών και των εγγύων. Πάντως, μα έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα, λέει η κυρία Βέσλοντ. Εδώ και δέκα χρόνια έχει αποδείξει η κυβέρνηση ότι δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντάλη, κύριε Επίτροπε. Απαντήσατε σε ένα πραγματικό μαραθώνιο ερωτήσεων, πολύ ουσιαστικά, πολύ ολοκληρωμένα μιλήσατε. Είδατε ότι σας χειροκροτούν θερμά, είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε μαζί σας, υπάρχει μεγάλη ε, επιθυμία εμπλοκής, είμαστε φιλόδοξοι, ε, θέλουμε να τηρούνται οι προθεσμίες όταν υπάρχουν στις νομοθετικές πράξεις και θέλουμε να εφαρμόζονται αυτά τα οποία αποφασίσαμε. Ευχαριστούμε και πάλι και εσάς και τους συναδέλφους σας, τους συνεργάτες σας. Θα σας δούμε και μια άλλη φορά στην Επιτροπή μας. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε λοιπόν Συνεχίζουμε λοιπόν με το θέμα υπαριθμών 16, καθολικός αριθμός και αριθμός εκτακτής ανάγκης 112. Η συγητής, ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με το 112 ως αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι καταλήλως ενημερωμένοι σε σχέση με αυτό τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Από την άλλη πλευρά μπορούμε επίσης να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι πολίτες ζητούν περισσότερες πληροφορίες και είναι διαθέσιμοι. Μόνο το 26% των πολιτών της Ένωσης μπορούν αυθόρμητα να ταυτίσουν τον αριθμό 112 με τον αριθμό που πρέπει να σχηματίσουν σε όλα τα κρατημέλη σε περίπτωση ανάγκης. Είναι μια μικρή πρόοδος της τάξης του 4% σε σχέση με το 2008. Μόνο το 35% θεωρεί ότι η πολίτες είναι καταλήλως ενημερωμένοι, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία, 96% θεωρεί πως είναι χρήσιμη η ύπαρξη του 112 του αριθμού έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο αριθμός θα πρέπει να είναι ένας αριθμός για όλους και οι πολίτες έτσι το εκλαμβάνουν και θεωρούν ότι το 87% των πολιτών ε, λένε ότι οι εθνικές αρχές οι αρμόδιες δηλαδή σε κάθε κράτος μέλος πρέπει και μπορούν να κάνουν περισσότερα για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε άτομα με ειδικέ ανάγκες. Είναι λοιπόν σαφές πως είναι απαραίτητη περισσότερη ενημέρωση, ε, δράσεις, ε, ευαισθητοποίησης και προτείνω αυτές τις δράσεις ευαισθητοποίησης στην έκθεσή μου. Δράσεις ευαισθητοποίησης που θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν από το σχολείο. Διαπιστώνεται ας πούμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη ότι η Ευρωπαϊκή ημέρα του 112 δεν ε, σηματοδοτήθηκε από καμιά πρωτοβουλία. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν, να ενημερώνουν και να προωθούν ε, ε, εκδηλώσεις σχετικές. Και είναι παράδεκτο να μην κάνουν τίποτα την Ευρωπαϊκή ημέρα του 112, στις 11 Φεβρουαρίου δηλαδή. Έχουμε την Ευρω... τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 που περιλαμβάνει πέντε στόχους ε, που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020 και όλα οδηγούν στο να πιστέψουμε ότι οι επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές για το επόμενο πολιετές πλαίσιο 2014 μέχρι 2020 θα πρέπει να οδηγήσει στο τουλάχιστον 85% των Ευρωπαίων πολιτών να μπορούν άμεσα και αυθόρμητα να ταυτίσουν το 112 ως τον αριθμό κλήσης έκτατης ανάγκης για όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί 80% γιατί πιστεύω ότι είναι ένας, ε, ένα νούμερο ε, που μπορεί να επιτευχθεί και θα πρέπει να υπάρχει ένας στόχος τέτοιος. Είναι βέβαια ανοιχτή, βέβαια ανοιχτό και στι απόψει των υπολείπων σε σχέση με αυτόν τον στόχο που θεωρώ ότι είναι εφικτός. Είναι επίσης πολύ σημαντική ο εντοπισμός μέσω δορυφόρου των κλήσεων. Όχι μόνο για να μπορέσει να βοηθηθεί αυτός που χρειάζεται βοήθεια, αλλά και για να αποθαρρυνθούν οι ε, ψευδείς κλήσεις. Γι' αυτό και θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει μια προσπάθεια από όλα τα κράτη-μέλη να συντονιστούν δηλαδή οι υπηρεσίες επικοινωνίας τους. Το 112 θα πρέπει να είναι μια υπηρεσία ποιότητας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει όντως να μπορεί να εντοπίζεται η κλήση για τους λόγους που σας προανέφερα. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρξει αυτή η υπηρεσία, όπως σας είπα, να είναι καθολική και οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από κάποια ειδική ανάγκη να μπορούν να το εντοπίσουν το νούμερο αυτό και να διευκολύνεται ε, η πρόσβαση για τα άτομα αυτά στον ε, νούμερο 112. Εξίσου σημαντικό είναι το θέμα της γλώσσας. Η γλώσσα να μην είναι εμπόδιο. για μια κλίση στο 112. Κάτι άλλο το οποίο δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση, αλλά εντωμεταξύ εγώ έχω παληθεύσει ότι γίνεται, είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα 112 αντίστροφο. Τι σημαίνει αυτό, και αυτό είναι δυνατόν, σε περίπτωση κάποιες επίγουσες ανάγκες, κάποιες καταστροφής, να είναι δυνατόν και μάλιστα είναι ευκταίο να συμβεί κάτι τέτοιο, να είναι τα παιδιά που θα, ε, τα παιδιά, οι άνθρωποι που θα κάνουν την κλίση να είναι η ίδια υπηρεσία που θα στέλνει ένα μήνυμα ή που θα κάνει κλήσεις ώστε να ενημερώσει για συγκεκριμένο κίνδυνο. Μπορεί να είναι μια χιονοστιβάδα, μια περνική καταστροφή ή να είναι σεισμός ή τσουνάμι όπως αυτό που έγινε στην Ιαπωνία. Οπότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακριβώς το 112 με την αντίστροφη όμως πορεία, ώστε να ε, έχει αυτή τη λειτουργία προστασίας, πολιτικής προστασίας. Τα κράτη-μέλη δηλαδή να είναι υπεύθυνα για να ενημερώσουν τον κόσμο για συγκεκριμένου κινδύνου. Γιατί ούτω ή άλλω ο βασικό μα στόχο είναι να προστατευτούν οι ανθρώπινε ζωέ και οι περιουσίε των ανθρώπων. Αυτές είναι οι προτάσεις που έχω συμπεριλάβει σε αυτήν την έκθεση. Και φυσικά είμαι ανοιχτό στις συμβολές των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. E, Ευχαριστώ συνάδελφε Φερνάντες, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα έχουμε κατάλογο μιλητών. Η κυρία Yes, Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση αυτή. Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Πρέπει το νούμερο αυτό να διαφημιστεί πολύ περισσότερο. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, τότε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν πρέπει να το θεωρούμε και τόσο δύσκολο. Κάθε ευρωβουλευτής σε κάθε ευκαιρία όταν απευθύνεται στα μέσα ενημέρωσης κάτι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει. Είναι σημαντικό νομίζω ο στόχος αυτός του 80% με τον οποίο συμφωνώ να προσπαθήσουμε να επιτευχθεί. Δεν έμαθα, δεν ήξερα για αυτό το νούμερο εγώ πριν γίνω ευρωβουλευτής, δεν ήξερα ότι υπάρχει, εκτός με, από ένα πολύ ασαφή τρόπο. Θέλω επίσης να συμφωνήσω και με την ιδέα του αντίστροφου 112. Πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε ίσως να συνεργαστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή για ε, όσα έκανε και προσβλέπω στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, η κυρία παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που ξαναδίνουμε προσοχή σε αυτό το 112. Είχα εμπλακεί στην υπόθεση πρόθεση του από το 2007 και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Με αυτή την εργαστία ευαισθητοποίησης ε, με τη δήλωση του Κοινοβουλίου κλπ. Καταφέραμε πολλά με κάποια επιτυχία, αλλά η γενικότερη επιτυχία του 112 είναι μάλλον περιορισμένη. 12 χρόνια και πάνω από τότε που δημιουργήθηκε είναι σχεδόν άγνωστο για ένα μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων. Ως εκπρόσωποι λοιπόν των πολιτών πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Το πρώτον, στο θέμα της ε, ευαισθητοποίησης. Είναι κρίσιμο. Γι' αυτό πρέπει να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο εισηγητής στην παράγραφο 3. Πρέπει διαρκώ η Επιτροπή να υπενθυμεί στα κράτη-μέλη ότι είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τους πολίτες ε, για το αριθμό αυτό και να παίξει ρόλο στην ενημερωτική εκστρατεία. Αυτό είναι ένα προφανές πρώτο βήμα δεδομένου τη βελτίωση των υπηρεσιών του 112 δεν θα χρησιμεύουν σε τίποτα αν τα τρία των πολιτών δεν έχουν ιδέα για την ύπαρξή του. Η υποχρέωση αυτή έχει επιβληθεί στα κράτη-μέλη εδώ και 9 χρόνια ήδη. Τα αποτελέσματα δεν είναι και εντυπωσιακά, πρέπει να παραδεχτούμε. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να αξιολογήσει αν τα κράτη-μέλη ε, ανταποκρίνονται παρκώ στις υποχρεώσει τους. Δεύτερον, το θέμα του ε, χρώματος. Ε, η επαρκής ενημέρωση για την τοποθεσία και το χρώμα μπορεί να ε, επιταχύνει τη διαδικασία και να σώσει ζωές. Επιπλέον από καιρού το θέμα των πληροφοριών αυτών για την τοποθεσία και το χρώμα ε, είναι μεγάλη, υπάρχει, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στην εφαρμογή και την αποτελεσματικά του μέτρου στα κράτη-μέλη. Πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ε, θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον αυτόματο εντοπισμό έχοντας υπόψη μας ότι θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να διατίθενται με κάποια ε, λογική καθυστέρηση λίγων ε, δευτερολέπτων. Αυτή η, ο εντοπισμός του, ε, του αυτού που κάνει την κλίση λοιπόν. Πρέπει Τέλος, να διαφημιστεί περισσότερο η ιδέα του αντίστροφου 112, ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των σε περιπτώσεις σοβαρών ε, επεισοδίων εκτάκτου ανάγκης. Θέλω απλώς να πω εδώ, πέρα από αυτά που ακούστηκαν, ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό. Μπορούμε να δείξουμε ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί αυτή η υπηρεσία στην οδηγία για την καθολική υπηρεσία πανευρωπαϊκή, πολυγλωσσή και διαθέσιμη σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και τώρα ο, ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μίλαν Καπέρνοκ, έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς. Ευχαριστώ. Αρχικά δεν είχα δει το λόγο, αλλά σας ευχαριστώ που τον δώσατε. Λοιπόν, ευχαριστώ τον εισηγητή. Εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα το γλωσσικό είναι και αυτό σημαντικό. Δεν αρκεί να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο 112, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος από την άλλη πλευρά να τους μιλήσει στη γλώσσα τους. Υπάρχουν εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας και θα τους άρεσε να υπάρχει ένας ε, που μιλάει τη γλώσσα τους. Επίσης, πρόσβαση από τον ε, χειριστή στις απαραίτητες ε, συμβουλές, τα απαραίτητα μέσα για να μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση για τα δικαιώματα των πολιτών για διαμεθοριακή περίθαλψη, συζητήσαμε τη δυνατότητα οι πληροφορίες υγείας να μπορούν να μεταδίδονται σε περιπτώσεις εκτάκτων ανάγκης. Οπότε και πάλι αυτή είναι μια περίπτωση που μπορούμε να το υπογραμμίσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα δεν ξέρω αν θέλει άλλος συνάδελφος το λόγο. Οπότε, ακούσουμε τον ε, πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι προτάσεις του εισηγητή και όλα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η Κομισιόν έχει σπίσει μια προτεραιότητα για τη διαθεσιμότητα και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του 112. Το 112 λειτουργεί και προσπαθούμε αυτό να πετύχουμε πάντα. Η γνώση για την ύπαρξή του βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική πτυχή. Αν όλα τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή ο εντοπισμός του καλούντος και η γλώσσα μπορεί να είναι άριστα, αλλά αν ο κόσμος δεν ξέρει ότι υπάρχει το νούμερο αυτό και δεν τηλεφωνάει, τότε τι να τα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Εμείς λοιπόν από πλευράς μας αποφασίσαμε να επιμείνουμε, ζητήθηκε εξάλλου από την Επιτροπή να ζητάμε από τα κράτη-μέλη να το γνωστοποιήσουν. Είναι κάτι που το κάνουμε διαρκώ με εμπειρογνώμονε, με ειδικού, με τα κράτη-μέλη, με την Επιτροπή επικοινωνία κλπ. Και, και συνεχώς του το υπενθυμίζουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε κατά νου να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Το θέμα είναι, αρκεί αυτό? Όχι προφανώς. Πράγματι, ο φιλόδοξος στόχος της ύπαρξης του ορίου 80% με το, μέχρι το 2020 μπορούμε και εμείς να τον προσυπογράψουμε από πλευράς μας. Τώρα, το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες ε, περιλαμβάνει διατάξεις για το 112, ήδη εθίγησαν η πρόσβαση σε αναπήρους χρήστες, ε, η δυνατότητα εντοπισμού του καλούντος, πολύ σημαντικό στοιχείο, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά την ε, μεταφορά της νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Κυρίως, όπως υπόθηκε, αυτό είναι η ακρίβεια και η ευθύνη του εντοπισμού του καλούντος ε, είναι θέμα του κράτους μέλους. Βεβαίω υπάρχει δυνατότητα να θεσπιστούν περαιτέρα μέτρα εναρμόνισης και να καθοδηγήσουμε το στοιχείο αυτό του εντοπισμού του καλούντος. Αυτή τη στιγμή ζητάμε από τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να κάνουν αυτά που πρέπει και αν χρειάζεται να μην διστάσουν να εισάγουν νέα μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα, για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και να βελτιώσουμε αυτή την έκθεση. Εγώ από πλευρά μου συμφωνώ με όλα όσα άκουσα. Πιστεύω λοιπόν πως θα καταφέρουμε να έχουμε μεγάλη συνένεση σε αυτόν τον στόχο, σε αυτή την έκθεση. Είμαι ανοιχτός και για άλλες προτάσεις, όπως είναι προφανώς, που θα φτάσουν, έχουμε χρόνο και για να καταθέσουμε τροπολογίες και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Και θα ήθελα να σας πω ακόμα ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θα λήξει στις 18 του μηνός Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 24 Μαΐου, στην ΕΜΚΟ στις 25 Μαΐου και στην Ολομέλεια με το καλό τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο θέμα τώρα. W tej chwili przerwa do godziny 17, dlatego że musimy po θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 5, γιατί πρέπει να περιμένουμε την κυρία Χάουκ, που είναι η σκιώδη συζητήτρια για το θέμα αυτό. Και της είπαμε να έρθει 5. Καλωσορίζω την κυρία Βαλτζάνη και περιμένουμε να έρθει η κυρία Χάουκ στις 5. Λοιπόν, αρχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι μετά το σύντομο αυτό διάλειμμα. Η για την Επιτροπή μας η συντάκτρια καλύτερα της γνωμοδότησης της Επιτροπής μας παρευρίσκεται όπως και η Γενική Εισηγήτρια του Κοινοβουλίου. Και περνάμε στο σημείο 17 εντολή για το τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012. Έχετε το λόγο, κυρία Βαλτάνη. Cari colleghi, la procedura di Αγαπητοί συνάδελφοι, η δημοσιονομική διαδικασία φτάνει σε μια σημαντική καμπή. Στις 20 Σεπτεμβρίου η Κομισιόν θα παρουσιάσει την πρότασή της για τον ε, προσωρινό προϋπολογισμό 2012 και το Κοινοβούλιο μας θα χρειαστεί να έχει μια ξεκάθαρη θέση κυρίως για να κατανοήσουμε πού ακριβώς θα πρέπει να ενεργήσουμε στους επόμενους ε, μήνες. Γιατί φέτος, όπως και πέρυσι, μια μόνο ανάγνωση του προϋπολογισμού επιβάλλει εξ αρχής σε όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η πρότασή μου για τον προϋπολογισμό 2012 την οποία συμμερίζονται καταρχήν οι συνάδελφοι της Επιτροπής Προπολογισμού και η Ολομέλεια είναι να βασιστεί ο προσωρινός προϋπολογισμός της Ένωσης με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Και άρα να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο που ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος, το 2011, και που είναι πραγματική δοκιμή συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, των, των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών και των προγραμμάτων μεταρρύθμισή του, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου οι μεταρρυθμίσεις και τη ίδια τη διακυβέρνηση. Η πρόταση λοιπόν λοιπόν είναι να γίνει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός το κλειδί του εξαμήνου για μια νέα ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, ούτως ώστε οι στόχοι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού να είναι σαφώς ορατοί, αναγνωρίσιμοι και να επιτρέπουν σύγκληση σε όλα αυτά των ε, πολιτικών των ε, μεμονωμένων ε, κρατών μελών που είναι όχι μόνο η προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία αλλά είναι και το μόνο σύστημα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε τις επενδύσεις που θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η κοινή στόχοι δεν μπορούν να είναι άλλη από την στατικική του 2020. Στόχοι φιλόδοξοι που πρέπει να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε άμεσα χωρίς να χάνουμε χρόνο γιατί η δεκαετία αυτή δεν μπορεί να μείνει με κενά σημεία δεν μπορεί θα πρέπει να είναι μια πολύ γεμάτη πορεία προς την επίτευξη των στόχων της επόμενης δεκαετίας. Αυτός ο προπολογισμό λοιπόν στην πρότασή μας θα ήθελα να είναι ένας προπολογισμό σύγκληση των προσπαθειών στους, με βάση τους στόχους της Ευρώπης για το 2020. Ένας προπολογισμό που βγαίνει από την Επιτροπή Προπολογισμών και θα να αποτελέσει σημαντικό θέμα για όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του Κοινοβουλίου που είναι οι μόνες που έχουν τις αρμοδιότητες και τις απαραίτητες γνώσεις για να μεταφράσουν σε συγκεκριμένο input τους στόχους της στρατηγικής 2020 ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Ε, Γι' αυτό και σιγά σιγά έχω έρθει σε ε, συνάντηση με όλες τις επιτροπές ε, ώστε να μπορέσουν να αγκαλιάσουν αυτό το θέμα του προπολογισμού σε ένα θέμα που αφορά όλες τις, προ... τις επιτροπές και όχι μόνο τον ε, προϋπολογισμό, την Επιτροπή Προϋπολογισμού και να μπορέσουμε να έχουμε ένα προφίλ για τις διάφορους τομείς μέσα στο μεγάλο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Ετούτη η Επιτροπή είναι αρμόδια για πάρα πάρα πολλά λεπτά ζητήματα που έχουν άμεση στέχη με δύο θεμελιώδεις στόχους της στρατηγικής, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, αλλά και έρευνα και ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχουμε δύο κλειδιά, σημαντικά θέματα επί των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πρωτοπόρος και όπου θα πρέπει τα επόμενα δέκα χρόνια να γίνουν μεγάλα βήματα πρόοδου. Καλό λοιπόν να αναζητηθούν από τώρα και να καθοριστούν ποιες από τις δράσεις, τα προγράμματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής θα είναι τα πιο στρατηγική σημασία για να μπορέσουμε άμεσα να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε εν ώψη τη στρατηγική 2020 με την άμεση προθεσμία τη 3η ε, Ιουνίου και που αφορά το προσωρινό κατάλογο πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων. Αυτά τα μέσα είναι πολύ ευαίσθητα γιατί επιτρέπουν στον προπολογισμό να γίνει ε, τροτός στις αλλαγές, στις ε, πετήσει ε, του κόσμου που μεταβάλλεται γύρω μα και άρα να προσαρμοστεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτά τα λεπτά λοιπόν προγράμματα θα παίρνουν ε, τμήμα των περιθωρίων μας και είναι απαραίτητο να προσέξουμε πάρα πολύ τα προγράμματα αυτά. Αυτό το χρόνο, εφόσον είμαστε στο τέλος της πραγματικής περίοδου που είναι αρμόδια γι' αυτό η κυρία η συνάδελφος Χάου κάνει μια πολύτιμη δουλειά στην Επιτροπή Σούρε και πλαισιώνουμε, ολοκληρώνουμε αυτό το πρόγραμμα δράσης με τον προπολογισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα άκαμπτος και ε, με πολύ στενά περιθώρια. Μας επιβάλλει δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλη φορά να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, σύντομοι στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και να συμμετέχουν όλα τα τμήματα που μας ενδιαφέρουν σε αυτό το σχέδιο του καθορισμού των στρατογικών προτεραιοτήτων. Και με ιδιαίτερη προσοχή βέβαια για τα προγράμματα, τα πιλωτικά και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. λαμβάνοντα υπόψη ότι από μια πρώτη έκθεση της Κομισιόν που αφορά αυτά που σήμερα είναι στον υπερπολογισμό απορρέει ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα σύμφωνα με την ε, Κομισιόν αλλά βέβαια θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα δεν είναι εφαρμοστέα και ή είναι εφαρμοστέα μετά από διάφορες άλλες ενέργειες. Να καταλάβουμε λοιπόν ποια προγράμματα λειτουργήσαν και ποια όχι και γιατί και να ξεκινήσουμε από αυτά που ήδη έχουν προταθεί και που έχουν λειτουργήσει σωστά. Η πρόσκλησή μου λοιπόν είναι αυτή, να να αναλυθούν ποιες δράσεις, ποια προγράμματα η αρμοδιότητα της Επιτροπής σας είναι ιδιαίτερα στρατηγική σημασία για την επίτευξη των στόχων στρατηγικής 2020 και να θεωρήσουμε αυτά τα προγράμματα ως γνώμονα για την δημοσιονομική διαδικασία ξεκινώντας από την ανάγνωση μετά την 20 η Απριλίου στον κατάλογο των προπαρασκευαστικών δράσεων και πιλωτικών προγραμμάτων αλλά και αργότερα ώστε να έχουμε ένα μέσο ανάγνωσης που θα πρέπει να κάνουμε όταν θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μας για τα νούμερα πλέον του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την συνάδελφο Φρανσέσκα Μπαλσάνη. Και τώρα θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια, τη συντάκτρια της δικής μας νομοδότησης εννοώ, την κυρία Γιώτα Χάουκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Φρανσέσκα που ήρθε ως εδώ Δύο φορές διατέλεσα γενική εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το Κοινοβούλιο και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ε, σκληρή δουλειά και πολλές επιτροπές θέλουν την εισηγήτρια να έρχεται να τους επισκέφτεται. Εμείς ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε σαφείς προτεραιότητες και ποια πράγματα θέλουμε να εφαρμοστούν. Πρώτο και κύριο βέβαια και προφανές είναι η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Και επίσης θεωρούμε ότι είναι εγκάρσια αυτή η υπόθεση και το καθήκον. Πολλά πράγματα που υπηρετούν την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι γνωστά και ξέρουμε ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα ε, το συγκεκριμένο κονδύλι του προπολογισμού κάθε φορά, αλλά θέλουμε να είναι εγκάρσια ε, η αρμοδιότητα αυτή και δεν ε, ενδείκνεται κανείς περισσότερο από τη Γενική Εισηγήτρια για να το πράξει αυτό. Και να κοιτάει σε όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού όπου θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να μπει αυτή η ιδέα της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής να το βάζει. Δεύτερον, βεβαίως και προφανώς το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για το περιβάλλον είναι το life στο περιβάλλον που πάει πολύ καλά πραγματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μεταξύ, οι υπηρεσίες δηλαδή, είναι σε θέση να εφαρμόζουν πολύ ωραία το πρόγραμμα LIFE. Τα κράτη-μέλη και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις τους κατάλαβαν πια πώς δουλεύει το σύστημα, ποια είναι τα σημαντικά μέτρα, ποια είναι τα σωστά μέτρα και επίσης το μέσο αυτό πρέπει να εξακολουθεί να ενισχύεται. Όχι μόνο στις σημερινές δημοσιονομικές προοπτικές, δηλαδή μέχρι το 2013, αλλά και πέρα από το 2013 θα πρέπει να συνεχιστεί για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή και πιο μικρών έργων, όχι με τα πολύ μεγάλα έργα, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τη βιοπικιλότητα, για τον αηφόρο βιώσιμο τουρισμό, όπως τα λένε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί το πρόγραμμα LIFE. Επίσης, ό,τι έχει να κάνει με την αποδοτικότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό από τα σημαντικότερα μέτρα που θέλουμε να εφαρμοστούν. Γνωρίζουμε ότι και η Επιτροπή Βιομηχανίας είναι βεβαίως αρμόδια, ενδεχομένως και η Περιφερειακή να είναι, διότι μέσω του μέσου συνοχής και τη διαρθρωτική πολιτική μπορεί να ασκήσει αυτή την πολιτική. Ωστόσο θα πρέπει να το πούμε αυτό και ω Επιτροπή Περιβάλλοντος και είναι για μα προτεραιότητα. Από πέρσι, το 2010, δεν έχουμε πια αρμοδιότητα ως Επιτροπή Περιβάλλοντος για την εκταμίευση πόρων για την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έχει μπει ε, στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ τώρα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθούνται και στα αναπτυσσόμενα κράτη τα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα δικά μας κριτήρια. Επίσης, πάντα θα πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι κάνουν αυτοί θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό με ναι, αυτά που θεωρούμε εμείς ε, αναπτυξιακή πολιτική με τη στενή ε, έννοια. Δηλαδή να μην κόψουμε από την ε, αναπτυξιακή βοήθεια για να τους πούμε ότι τώρα πάρτε αυτά τα χρήματα για το κλίμα. Και τέλος, χωρίς αυτό να είναι λιγότερο σημαντικό, η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία του κλίματος είναι τριπλή υπόθεση. Συνεργασία με τα κρατη συνεργασία από τον προπολογισμό με κίνητρα, αλλά κυρίως και πάρα πολύ σημαντικό με την νομοθεσία. Είναι τριπλή προσπάθεια. Και αφού συζητούμε για την νομοθεσία, θα πρέπει και πάλι να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι εντάξει καλή νομοθεσία, θα πρέπει να ελέγχουμε και την εφαρμογή της. Επιγόντως χρειάζεται αυτός ο έλεγχος. πώς να το πω, μπορούμε να κοιτάμε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς έχει προσφύγει επί παραλήψη. Είναι 2.362 από τις οποίες ε, υποθέσεις, 419 δηλαδή 17% αφορούν την παραβίαση της νομοθεσίας για το περιβάλλον από όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο δικαστήριο. Ε, αυτό μπορεί να το επομιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους εργαζόμενους στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αρκεί το προσωπικό. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καμιά φορά είναι επιφυλακτική όταν ζητάει προσωπικό, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε αν μπορούν, τους καλύπτει αυτό, υπάρχει έλλειψη προσωπικού ή όχι. Και μπορούμε να ασκήσουμε αρκετή πίεση στα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν κατά αυτόν τον τρόπο την νομοθεσία. Με ενδιαφέρει. Και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει. Και δεν με ενδιαφέρει μόνο ως εισηγήτρια για τον προπολογισμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά γενικότερα και ως πρόεδρο αυτό τον καιρό της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ, ξέρετε, της έκτακτης Επιτροπής που ασχολείται με την εξασφάλιση των πόρων μετά το 2013. Γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση όπου θα ασχοληθούμε με την διοίκηση. Εκεί θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται με το προσωπικό. Αν μα έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να βάλει και το χέρι στην τσέπη. Ξέρω ότι δεν είναι δημοφιλές να λέμε θέλουμε περισσότερο προσωπικό. Εντάξει, εξίσου δημοφιλές είναι να βλέπουμε σε ορισμένα κράτη-μέλη να μην τηρείται η ε, νομοθεσία για το περιβάλλον, να μην εφαρμόζεται και αν δούμε ακριβώς ποιες είναι οι διαδικασίες προσφυγής επί στο δικαστήριο, αυτά σωρεύονται ε, σε μερικά κράτη-μέλη. Άρα χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε και να θέλουμε απάντηση. Αν μπορείτε να μας απαντήσετε ακόμα καλύτερα. Αν δεν μπορείτε τώρα, θα σας παρακαλούσα μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή δυνατόν στην έκτακτη συνεδρίαση. Όχι, συγγνώμη, διορθώνει η κυρία Χάουκ. Δεν είναι την άλλη εβδομάδα η συνεδρίαση τη Επιτροπή Σούρε, είναι μετά το Πάσχα. Αλλά δεν πειράζει. Θα ήθελα κάποια στοιχεία από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το προσωπικό, για να το δούμε και με τον αρμόδιο επίτροπο για τη διοίκηση και να τα συζητήσουμε στην Επιτροπή Σούρε και να προβάλλουμε και τα αιτήματά μα. Ένα τελευταίο. Είναι μάλλον έκκληση αυτό σε όλου του σκιώδει ηγητέ και όσους ενδιαφέρονται στις πολιτικές τους ομάδες και είναι αρμόδιες, αρμόδιοι. Έκκληση να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Είπε η Φραντσέσκα ότι στις 3 του Ιούνιου λίγη προσωρινά η προθεσμία για την κατάθεση καλών ιδεών και εμείς έχουμε εσωτερική διαβούλευση και εσωτερικό χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και θέλουμε να κοιτάξουμε με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει και υλοποιεί αυτά που αποφασίσαμε πέρσι για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και δεν μπορώ παρά να συμβουλεύσω και να παρακινήσω όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται και έχουν κάνει καλές προτάσεις να έρθουν αύριο στην Επιτροπή Προϋπολογισμού 9 με 11 έχουμε ακρόαση ακριβώς για αυτά τα θέματα. Γνωρίζω ότι η Εμίλια που είναι πραγματικά το μαργαριτάρι της ε, Επιτροπής μας για τον προϋπολογισμό ξέρω ότι το έχει στείλει σε όλες τις πολιτικές ομάδες αλλά δεν πειράζει να το επαναλάβουμε και εδώ. Είστε όλοι προσκεκλημένοι να έρθετε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και να ακούσετε τι είναι τα πιλωτικά προγράμματα, τι μπορούν να επιτύχουν και πώς θα πρέπει να είναι φτιαγμένες έτσι οι ιδέες ώστε να αναγνωριστούν ως πιλωτικά προγράμματα, πώς θα πρέπει να είναι πλεγμένες ή κεντυμένες στην κατασκευή τους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, την κυρία Γιούτα Χάουγκ. Και τώρα, επόμενος ομιλητή στον κατάλογο μου. Ποιος είναι? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω μιλώντας βουλγάρικα, λέει ο κύριος Παναγιώτοφ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάουγκ για τη δουλειά της και να τονίσω επίσης ότι κατά την άποψή μου η κυρία χάουγ ε, ανήκει στις ηγετικές φυσιογνωμίες του Κοινοβουλίου μας. Την ευχαριστώ πολύ. Ως σκιώδης εισηγητής θα ήθελα να τονίσω το εξή. Το χρονοδιάγραμμα, το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ανταλλαγή απόψεων και την τελική προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών είναι πάρα πολύ βραχή. Και θα ήθελα να ρωτήσω δεν θα ήταν πιο σκόπιμο να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Επιτροπή μας καλύτερα μεγαλύτερη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και να βάλουμε τελική προθεσμία αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό τον καιρό αναλύω εγώ την αποτελεσματικότητα του προϋπολογισμού του 2010 και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η αρχή της χρηστής ε, εκτέλεσης του προπολογισμού. Διαπιστώνουμε μια τάση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάει πιο πολύ τα ε, αριθμητικά στοιχεία, τα ποσά και όχι τα πραγματικά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό για το 2012 λοιπόν, θα ήθελα περισσότερους πόρους ε, για το περιβάλλον και για προγράμματα μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Συγκεκριμένα μέτρα για ενεργειακή απόδοση, πρόθεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, αξιοποίηση των καυσίμων και κυρίως των σπανιών καυσίμων στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την κρίση στην Ιαπωνία, πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, στην Επιτροπή μας, οπωσδήποτε. Θα γίνουν αντίστοιχες προτάσεις για τα πιλωτικά προγράμματα, για την ενεργειακή απόδοση και την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πολιτήμων πρώτων υλών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και την κυρία Χάουκ άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιώτοφ. Αν δεν θέλει κανένας άλλος ε, συνάδελφος το λόγο, τότε... τότε υπάρχει παρίστατο ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγγνώμη. Euh, Μήπως η, η, η θα ήθελε και πάρει το λόγο. Όχι. Πολύ σύντομα. Να απαντήσω στη συνάδελφα. Ευχαριστώ για τις ε, υποδείξεις αυτές που συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική 2020 κατά πολέμηση των κλιματικών αλλαγών, ενεργειακή επάρκεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναμφίβολα είναι από τις σημαντικότερα στοιχεία της στρατηγικής 2020 και δυστυχώς είδαμε ότι υπάρχουν ε, ε, και εδώ προβλήματα και πρέπει να πιέσουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα. Επίση, να ευχαριστήσω για την αναφορά που έκανε η Γιούτα Χάουγκ για την επίβλεψη τη εφαρμογή τη νομοθεσία. Είναι αυτή η προστεθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Γιατί θύμιζα ότι πρόκειται και για τι μεταρρυθμίσει. Δηλαδή, ο συντονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εθνικά κράτη θα πρέπει να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στον προπολογισμό, για να φτάσουμε και σε συντονισμό, το κρίσιμο συντονισμό των νομοθεσιών. Η διορία για τα πιλωτικά προγράμματα προγράμματα και τις προσφυγικες δράση δράσεις είναι Ιουνίου και συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να έχουμε ένα feedback από την Κομισιόν. Είναι μια διορία για μια προσωρινή πρόταση, γιατί στη συνέχεια από την τεχνική άποψη αυτό το προγράμματα και οι δράσει αυτέ είναι πραγματικέ τροπολογίε για τον προπολογισμό. Θα έχουμε δηλαδή επίσημη προθεσμία για το Σεπτέμβριο. Αλλά για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα δημιουργηθούν ε, σκοτεινά αποθεματικά, δηλαδή να κάνουμε ε, ε, φτιάξουμε κονδύλια τα οποία μετά να μην μπορεί να τα εκτελέσει η Κομισιόν. Ε, θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση Κομισιόν στην Κομισιόν, να κάνουμε μια πρώτη πρόταση στην Κομισιόν για να δούμε πώς θα βλέπει εκείνη και μετά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο συγκεκριμένα και πιο αποτελεσματικά επειδή, όπως σας είπα, τα περιθώρια είναι πολύ πολύ μικρά. κυρία Χάουκ, ευχαριστώ. Θέλω να υπογραμμίσω αυτό το τελευταίο. Γιατί ό,τι αποφασίζουμε εμείς στον προπολογισμό και στη συνέχεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί, είναι λεφτά που πάνε στο βρόντο. Εμείς τα χάνουμε. Δεν μπορούμε κατά τη διάρκεια του έτους να κάνουμε καμιά μεταφορά πιστώσεων, επαναγραφή στον προϋπολογισμό. Στις 31 Δεκεμβρίου γυρνάει στο κρατικό κορβανά, στο Υπουργείο Οικονομικό κάθε χώρας. Δεν το θέλουμε αυτό και δεν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Όπως κάθε χρόνο, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ πέρα, ε, φωνάζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τι είναι πιλωτικό πρόγραμμα, τι μπορεί να είναι προπαρασκευαστική δράση, πώς θα πρέπει να αναπτύσσεται, ενδεχομένως πριν το υποβάλουμε ε, μπορούμε και πριν το αποφασίσει η Επιτροπή μας να το έχουμε κοιτάξει και συζητήσει με κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρωτήσουμε εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Έχει ελπίδες να ευδοκιμήσει, να εφαρμοστεί. Μην χάσουμε τα λεφτά. Γιατί κάθε φορά που έχουμε μια λεγόμενη έτσι, νομοθετική βάση ή νομική βάση, εν πάση περιπτώσει, τεχνικό όρο, αυτό, σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι έχει χαθεί από πιλωτικό πρόγραμμα. Τα πιλωτικά προγράμματα είναι καινοτόμε ιδέε, φρέσκα μέτρα, καινούρια που εμεί προτείνουμε ω κοινοβούλιο. Αλλά να είναι πραγματικά ολοκένουρια, να μην έχουν ξανακουστεί πουθενά, χωρί νομική βάση, χωρί άλλα προγράμματα ή λοιπά που έχουμε. Το ξέρω ότι είναι δυσκολία και κάθε χρόνο δυσκολεύει ακόμα και περισσότερο η κατάσταση, θα πρέπει να το καταλάβουμε γιατί και ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε όλο και πιο ολοκληρωμένοι και έχουμε περισσότερη νομοθεσία και πιο πολλές νομικές βάσεις για όλα αυτά που κάνουμε. Παρ' όλα αυτά σίγουρα υπάρχουν τομείς και καλές ιδέες που δεν έχουν νομική βάση και μπορούν να υποβληθούν για τον προπολογισμό, αλλά παρακαλώ όχι σπατάλη. Τελεία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και με αυτή την έκκληση της κυρίας Χάουκ ε, προς τη φαντασία μας, ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Θέλω να σας πω μόνο ότι μπορείτε να κάνετε τροπολογίες μέχρι τις 15 Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 8 Σεπτεμβρίου και τα πιλωτικά προγράμματα και τα λοιπά μπορείτε να τα υποβάλλετε ως ιδέες στη γραμματεία το αργότερο μέχρι τις 25 Μαΐου. Γιατί τότε θα συζητήσουμε αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Μέχρι τις 15 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι σας είπα είναι οι τροπολογίες για το σχέδιο προϋπολογισμού. Λοιπόν, αυτά. Τελειώνει και αυτό το σημείο όπως και η συνεδρίαση της Επιτροπής και ακολουθούν αμέσως οι συντονιστέ. Ευχαριστώ πολύ.